Καλό απόγευμα συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας σε αυτήν την θητεία. Ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι ήδη έχουν ξεκινήσει την εκστρατεία τους, αλλά ξέρω ότι και άλλοι θα έρθουν να μας βρουν σήμερα το απόγευμα. Σημείο 1. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να εγκρίνουμε το σχεδίο της ημερησίας διατάξεως. Δεύτερο σημείο ανακοινώσεις Πρόεδρου. Καταρχάς τα καλά νέα. Την περασμένη εβδομάδα εγκρίναμε το νέο μέσο ανάπτυξης σε πρώτη ανάγνωση Στρασβούργο με σημαντική πλειοψηφία καμία από τις προτάσεις τροπολογίας δεν εκρίθη, Έχουμε λοιπόν τελική θέση αυτή που είχαμε εγκρίνει, δηλαδή εμείς και η ΑΦΕΤ. Τι θα γίνει μετά, ό,τι μαντέψει ο καθένας. Το Συμβούλιο διαμορφώνει εγώ τη θέση του. Τα πράγματα είναι αβέβαια, γιατί έχουμε το θέμα του EDF, ε, του προϋπολογισμού κτλ. Όλα αυτά θα εισέλθουν στη συζήτηση για το μελλοντικό πιδριελταπή. Τι σημαίνουν αυτά για μας, ότι ο φάκελος θα παραδοθεί στην επόμενη σύνθεση. Οι συνεισηγητές θα πρέπει να αναδιοριστούν ή να οριστούν από την αρχή. Θα μπορούσε αυτό να γίνει πριν από τη θερινή διακοπή ή όχι και να ξεκινήσουν τριμερείς διάλογοι ή όχι ανάλογα με τη θέση του Συμβουλίου. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους και την γραμματεία γιατί ήταν σκληρή η δουλειά και περίπλοκη. Τώρα, οι ημέρες της ανάπτυξης 18 και 19 Ιουνίου για να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες και να αναπτύξουμε μια κοινωνία στην οποία κανείς δεν θα ξεχνιέται, δεν θα αφήνουμε κανέναν πίσω, έξω. Έχουμε τα μέλη του Κοινοβουλίου που όλοι συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών θα είναι μέλη. Θα χρειάζονται για την εκδήλωση κάποια μπάτζ, παρακαλώ ελάτε σε επαφή με την γραμματεία αν επιθυμείτε να προσέλθετε. Στις ημέρες αυτές της ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν έχω άλλες ανακοινώσεις. Ίσως να έχουμε κοινή συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα με την ΑΦΕΤ για να ακούσουμε για τελευταία φορά την κυρία Μαγκερίνη στο Στρασβούργο. Οι συνάλληφοι θα το συζητήσουν απόψε για να συζητήσουν για την παγκόσμια στρατηγική, ώστε να είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν την ολοκλήρωση της Έχουμε τα πρακτικά της 21ης-22ης Ιανουαρίου, 27 Φεβρουαρίου, όλα αυτά είναι στα, στους φακέλους σας. Αν έχετε σχόλια, παρακαλώ να τα δώσετε στη γραμματεία πριν το τέλος συνεδρίασης. Ιδάλλως θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί. Σημείο 4. Ανακοινώσει τη Επιτροπή. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή έχει κάποιε ανακοινώσει για μα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, γιατί αναφερθήκατε στι δύο ανακοινώσει, αλλά είχαμε κάποιε καθυστερήσει. Η στρατηγική τη Νοτιού Αμερική θα υιοθετηθεί μέσα Απριλίου και τη κεντρική Ασία μέσα Μαΐου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Η γραμματεία είμαι σίγουρη ότι σημείωσε. Νομίζω ότι ήταν στο planning του 17 ήδη αυτά που είπατε, τέλος πάντων. Έστω και αργά έρχονται τώρα. Άλλες ανακοινώσεις δεν έχουμε από την Επιτροπή, ευχαριστώ. Ώρα των ερωτήσεων δεν έχω λάβει ερωτήσει για τη συνεδρίαση. Πάω στο 6. Συζήτηση για, την, ε, για το φόρουμ υψηλού επίπεδου του των Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε εδώ τους συναδέλφους για να μας μιλήσουν για το τι τρέχει, τι συμβαίνει με τις προπαρασκευές του, για το φόρουμ του Ιουλίου και το υψηλού επίπεδου, πώς να το πω, τη σύνοδο κορυφής. Θα έχουμε φόρουμ υψηλού επίπεδου και το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων για πρώτη φορά το 2015 θα επανεξετάσουν πού βρισκόμαστε με τους στόχους βιωσίμου ανάπτυξης. Και θα υπάρξει, θα προσιαστεί και μια συνολική εικόνα για το πώς τα πάει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους στόχους βιωσίμου ανάπτυξης. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη, εκτός ίσως από ένα ή δύο, παρουσίασαν τις σχετικές δικές τους απόψεις και πρέπει να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, συνεργασία για την ανάπτυξη που η ΔΕΒΚΟ προετοιμάζει και πώς αυτό συνδυάζεται με το έγγραφο ανάλυσης. Το Κοινοβούλιο ήδη ψήφισε το Μάρτιο. Ε, ταχθήκαμε υπέρ της επιλογής 1 λοιπόν μεταξύ των επιλογών αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε για το πώς προετοιμάζεστε για τις δύο αυτές εκδηλώσεις και ίσως διευθυνίστε μας είναι τον Ιούλιο ή το Σεπτέμβριο που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσει συνθετικά τη δική της θέση. Θα υπάρξει εξοδότηση από την Επιτροπή μας, ε, ε αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη και το Σεπτέμβριο κοινή αντιπροσωπεία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και ίσως με άλλες. Ποιο θα πάει και πώ θα γίνουν όλα αυτά και πώ θα διοργανωθούν, θα συζητηθούν αυτά μετά τι ευρωπαϊκέ εκλογέ, Δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Um, Ευχαριστούμε πολύ Λίντα. Καλό απόγευμα σε όλους και όλους. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας για το πού βρίσκεται η προπαρασκευή του HPF και για την έκθεση, για την Joint Synthesis Report. Τώρα, δύο πράγματα. Πρώτα, να ρωτήσω πόση ώρα μου δίνετε χρόνο. Έχετε, έχετε χρόνο. Έχουμε, έχουμε χρόνο. Πολύ ωραία. Αρχίζω λοιπόν με την Joint Synthesis Report. Όσο γνωρίζετε, στην ε, συνένεση έχουμε ε, γραμμένη την υποχρέωση για την έκδοση της έκθεσης. Κάθε τέσσερα χρόνια. Ε, ξεκινώντας από φέτος. Και μετά ανά τετραετία όταν το HPF ανεβαίνει σε ένα επόμενο επίπεδο. Έκθεση λοιπόν για τα πεπραγμένα. Έχουμε συντάξει την έκθεση αυτή με τρόπο συμμετοχικό μαζί με τις χώρες μέλη. Γιατί η ιδέα πίσω από την έκθεση είναι να δείξουμε τι κάνουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και τι κάνουν από κοινού οι χώρες μέλη. Ήμασταν σε επαφή και μαζί σας, διαβάσαμε και τη δική σας έκθεση και έχουμε περιλάβει και ε, τα όσα επιθυμείτε κι εσείς ε, στο σχέδιό μας που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε την joint σύνθεση report τον Απρίλιο, ώστε το Συμβούλιο να έχει χρόνο να την εξετάσει και εμείς να μπορέσουμε να ε, παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα τον Ιούλιο και όχι τον Σεπτέμβριο όπως είπα στην αρχή εκ παραδρομής. Όταν θα έχουμε ολοκληρώσει την εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως σε ορισμένα σημαντικά θέματα που είναι και κάπως οριζόντια μέσα στην συνένεση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το θεματολόγιο το οποίο διασυνδέεται και πού βλέπουμε ε, βελτιώσεις ή πού βλέπουμε αναγκαίες βελτιώσεις. Για την ώρα η έκθεση βρίσκεται στο στάδιο της συντάξεως. Να σας δώσω κάποιες ιδέες για το ποια πράγματα βλέπουμε να εμφανίζονται ως βασικά ζητήματα του περιεχομένου της. Μπορούμε να πούμε συνολικά ότι οι χώρες μέλη των, του ΟΗΕ κάνουν πολλά πράγματα σε μεγάλο αριθμό χωρών. Έχουμε λοιπόν θετικά μηνύματα και είναι σημαντικό να τα πούμε. Η έκθεση θα λέει ότι γίνεται πρόοδος για βελτιωμένη συνεργασία με τις χώρες μέλη, πώς έγινε στο παρελθόν, κοινό προγραμματισμός για την εφαρμογή επίσης, πώς διασυνδέονται οι στόχοι, πώς ενσωματώνονται στην, στο θεματολόγιο ανάπτυξης τα διάφορα θέματα, πώς ε, λαμβάνουμε υπόψη την, ε, τα, τη μεγάλη φτώχεια, ζητήματα ανισότητας, προώθησης της ειρήνης και σταθερότητας, επίσης τι κάνουμε για τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει για την αναπτυξιακή βοήθεια, πώς προσπαθούμε να φτιάξουμε έτσι την συμμετοχή μας να είναι κομμένη και ραμμένη τις ανάγκες των συμμετοχουσών χωρών και πώς συντονιζόμαστε με άλλους εταίρου στην αναπτυξιακή βοήθεια όπω τα Ηνωμένα Έθνη. Θα μπορέσουμε να δείξουμε λοιπόν τα θετικά αυτά σημεία της προσπάθειάς μας, ελπίζω. Τίποτα βέβαια δεν είναι τέλειο και θα τονίσει η έκθεση και ορισμένους τομείς όπου πρέπει να γίνει η εντονότερη προσπάθεια στο μέλλον. Θα έρθουμε σε αυτά. Νομίζω ότι ορισμένοι από τους τομείς όπου πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο στο μέλλον είναι η στενότερη ευθυγράμμιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την Ατζέντα 2030. Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη διαδικασία, σαφώς. Εμείς δηλαδή και οι χώρες μέλη προσαρμόζουμε το σύστημά μας στις νέες ανάγκες θα πρέπει να γίνει πιο πολύ όμω στο μέλλον αυτό. Συνεργαζόμαστε, όπως είπα, με τις χώρες μέλη στα πλαίσια σεναρίων θα μας επιτρέψουν να προοδεύσουμε και στο μέλλον. Το είπα αυτό. Η ιδέα ότι πρέπει να διαρθρωθεί ο διάλογος με τις χώρες εταίρους και για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και σύμφωνα και με τα δικά τους προγράμματα για να δούμε πώς η συνεργασία μπορεί να ενταχθεί στη συνολική αυτή προσπάθεια. Και να προσαρμόζουμε βέβαια τη συλλογή δεδομένων και ανάλυση στις, στις νέες ανάγκες των ε, ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αναμένουμε και θα θέλαμε η έκθεση να είναι στέρεα, σύντομη, στοχευμένη και εύκολο να παρουσιαστεί στο κοινό επικοινωνιακά. Αυτό προσπαθήσουμε να κάνουμε. Η δομή θα είναι τη τάξη των 15 σελίδων η δομή της έκθεσης. Με τα ουσιώδη των όσων κάνουμε, σύμφωνα και με τα πέντε κεφάλαια της Ατζέντα 2030 και μετά σε παράρτημα διάφορα δελτία ή επιμέρου θέματα. Από στόχους βιώσιμη ανάπτυξη 1 έως 17. Πρώτη φορά συντάσσουμε τέτοια έκθεση. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε. Με τα στατιστικά εργαλεία που διαθέτουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα περιλάβουμε και πολλά παραδείγματα. Είναι βέβαια το πρώτο βήμα και ελπίζουμε να βελτιωθούμε στο μέλλον, ώστε στην επόμενη έκθεση να μπορέσουμε να την κάνουμε πιο στοχευμένη ακόμη. Και ελπίζουμε επίσης ότι αυτή η κοινή έκθεση με τις χώρες μέλη από μόνη της θα μπορέσει να αποτελέσει ένα μηχανισμό που να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε περαιτέρω με τις χώρες μέλη. θα παρουσιαστεί στην HLPF στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο. Η υπόθεση στην οποία βασιζόμαστε τώρα είναι να την υποβάλουμε σε ένα side event που θα δείξει τη συνολική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή του θεματολογίου 2030 και εσωτερικά και εξωτερικά. για τους στόχους, για, τον, για το κείμενο προβληματισμού που έχει διεγκριθεί για την έκθεση της Ευρωστάτ που θα δημοσιευθεί επίσης τον Ιούλιο και με την έκθεση PCD που έχετε ήδη δει. Αυτές είναι οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν για τη σύνταξη της έκθεσής μας. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, εμείς Έχουμε πάρει το περιεχόμενο που βλέπουμε για τις εξωτερικές πτυχές του εγγράφου προβληματισμού που προβλέπει και τις τρεις επιλογές. Και κάθε από αυτά θα βασίζεται στην εφαρμογή της συνένεσης στην πραγματικότητα και περισσότερο για τις εξωτερικές πτυχές που θα είναι μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας. Πάλι για το HLPF είναι σημαντικό νομίζω να παρουσιάσουμε εκεί την έκθεση διότι φέτος το HLPF έχει μεγάλη σημασία. Και δύσκολο κατά κάποιο τρόπο. Πρώτα, διότι πρόκειται για το τέλος ενός κύκλου. Ενός κύκλου τεσσάρων ετών, που θα πρέπει να δούμε αν βρισκόμαστε στη σωστή πορεία και τι να κάνουμε στο μέλλον. Και το Σεπτέμβριο αρχίζουμε την επανεξέταση του HLPF. Δεύτερο, είναι σαφές ότι για κάποια μέρη του θεματολογίου αυτά αμφισβητούνται από κάποιους από τους εταίρους και δεν είναι απολύτω ε, μέσα στην προσπάθεια και αυτή. Άρα πρέπει να τα προστατεύσουμε τα τμήματα αυτά του θεματολογίου. Άρα πρέπει να εξηγήσουμε ακριβώς τι και γιατί το κάνουμε. Είπα λοιπόν παρουσίαση σε υπουργικό επίπεδο τον Ιούλιο, που θα γίνει και επανεξέταση ενός αριθμού στόχων, καθώς και οι εθνικές εθελοντικές επανεξετάσεις. Θα συμμετάσχουμε ως συνήθως στην διαδικασία των επανεξετάσεων, review. Οι στόχοι που θα συζητηθούν είναι για την παιδεία, κλίμα, ειρηνικές και σταθερές κοινωνίες και η σχετική εφαρμογή θα γίνει και πολιτική διακήρυξη, αλλά μία, που θα εγκριθεί τον Σεπτέμβριο. Αλλά οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν τώρα. Και τη διευκόλυνση κάνουν εκεί Μπαχάμες και Σουηδία. Θα είναι σημαντική διακήρυξη αυτή. Θα πρέπει να αποφύγουμε να γίνει μια ευκαιρία για ξύλωμα του θεματολογίου. Σημειώνουμε ότι πέρσι οι Ηνωμένε Πολιτείε κατεψήφισαν το ψήφισμα. Εκεί έχουμε ένα θέμα. Ο σωστός δρόμος, κατά τη γνώμη μας, είναι να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια σύντομη, στοχευμένη πολιτική διακήρυξη που να μην ξανανοίξει το θεματολόγιο, αλλά να στοχεύσει στο πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την επιτάχυνση στο μέλλον. Να δώσουμε δηλαδή μια θετική όθηση σε ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε. Και θα συνεργαστούμε μαζί σας και με τις χώρες μέλη και με άλλους που έχουν την ίδια προσέγγιση. Να αρκεστώ λοιπόν σε αυτά και ευχαρίστως να σας απαντήσω αν έχετε ερωτήσεις. Η πρόεδρο. σα ευχαριστώ. Έχω ερωτήσει. ξέρω όμω ότι θέλετε να μιλήσει και η συνάδελφό σα, Η κυρία Ντεμπέργκα από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, που ίσω να μας εξηγήσει τον ρόλο της υπηρεσία της. Εσείς ε, ασχολείστε περισσότερο με την πολιτική διπλωματία. Και εγώ ανησυχώ διότι ενδέχεται να ανοίξει ξανά το θεματολογίο από την αρχή και νομίζω πέρσι η Πρέσβηση των Ηνωμένων Εθνών είχε πει ότι θα επανεξετάσει ολόκληρη διαδικασία. Τι ακούμε για την ε, στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστώ και καλό σας απόγευμα σε όλους και όλους. Σχετικά με το δικό μας ρόλο τώρα, συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και DEFCON προκειμένου. με παρόμοιες αναλύσεις για τα διακυβευόμενα και τώρα 2019 είναι σημαντικό να ε, δώσουμε νέα πνοή στο θεματολόγιο για τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία του HLPF του Ιουλίου καθώς και την ε, διάσκεψη του Σεπτεμβρίου γιατί είναι και ζήτημα αξιοπιστία για την πολυμερή ε, προσέγγιση και για τη διεθνή κοινότητα γενικότερα για να δείξει ότι αυτή η πολυμερής αντιμετώπιση των προβλημάτων προσφέρει ωφέλη στους πολίτες. για την εφαρμογή των SDG, των ε, στόχων βιώσιμη ανάπτυξη, είναι και ζήτημα αξιοπιστία. Όπω το βλέπουμε από την σκοπιά τη υπηρεσία μα. Και βέβαια για να εφαρμοστεί η συνολική στρατηγική της Ένωσης, όπου είναι ένα σημαντικό οριζόντιο στοιχείο η στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σύνταξη της εκθέσεως για στήριξη των Ηνωμένων για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης έγκαιρα ώστε να τονιστεί και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην HLPF για να γίνει αυτή επιτυχία. Τονίζω επίσης και πάλι την σημασία της ευκαιρίας αυτής για να τονιστεί η πρόοδος αλλά και η δουλειά που μένει να γίνει ακόμη με καλύτερη συνεργασία και ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ως χώρες με κοινό προγραμματισμό και κοινή εφαρμογή αποφάσεων. Να δείξουμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε διότι θεωρούμε ότι είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος αυτός για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή και μια ενιαία φωνή της Ένωσης και σε επίπεδο κρατών. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή που ανοίγεται και επίση να συνεργαστούμε ακόμη στενότερα και επί τόπου και τον ε, εκ νέου ενισχυμένο ρόλο των συντονιστών και να ενισχύσουμε και τις προσπάθειες των ε, εταίρων χωρών για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με συμμετοχή των ε, συντονιστών που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες αυτές. Να με επιτρέψετε και εμένα να αρκεστώ σε αυτά και να παρακολουθήσω την υπόλοιπη συζήτηση. Ευχαριστώ. Εδώ έχουμε τον ειδικό για θέματα ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Εγώ Ευρωβουλευτής είμαι, αλλά αυτά τα θέματα με ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. Όποτε, από τότε που ξεκίνησε το έτος της ανάπτυξης μετά την, τις εκλογές, νομίζω ότι έχουν υπάρξει κάποιες πολύ σημαντικές επαναστατικές ευκαιρίες. Γενικώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Η υπηρεσία σας ε, εντός της Κομισιόν πιέζει πάρα πολύ Και από ό,τι ξέρω, θυμάμαι πολλές φορές να έχω ε, ε, καθίσει μαζί με την ε, Φεντερίκα Μογκερίνη, τον κύριο Νίμιτσα, τον Φραντ Τίμερμαν στη Νέα Υόρκη για, τις, για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και πώς μπορούμε να τα προωθήσουμε. Πολλές φορές δεν είμαστε εκεί που πρέπει, εκεί που νομίζαμε ότι θα έπρεπε. Η Κομισιόν η ίδια δεν έχει βέβαια αποκλείσει το τι θα μπορούσε να γίνει. Ωστόσο, το κοινοβούλιο δεν είναι, για το κοινοβούλιο δεν είναι ξεκάθαρο ότι έχουν ε, εκφραστεί πλήρως όλοι οι στόχοι της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχουν πάρα πολύ, σημαντικοί, πάρα πολύ σημαντικές πτυχές όπως ε, ε, το εμπόριο, τα οικονομικά θέματα, ε, στα οποία ακόμα πρέπει να υπάρξει πρόοδος. Οπότε δεν καταλαβαίνω γενικώ πώς θα μπορούσε να έχει παρέμβει περισσότερο το Κοινοβούλιο. Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές ε, προέρχονται από θέματα που άπτονται της πολιτικής ανάπτυξης, από τομείς που άπτονται της ε, πολιτικής ανάπτυξης. Και νομίζω ότι ε, έχουμε βέβαια προχωρήσει αρκετά και από την πλευρά των κρατών μελών, αλλά χαίρομαι που εδώ στο Κοινοβούλιο ακούμε ε, ότι η Φιλανδία, μια σκανδιναβική χώρα, είναι ένα υπόδειγμα ότι τα πράγματα όντως προχωρούν. Ερώτημα λοιπόν. Σε αυτή την έκθεση Λέτε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεκτική συζήτηση. Υπάρχουν κράτη-μέλη που όντως έχουν φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο και να έχουμε ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια καλά παραδείγματα από τα 28 κράτη-μέλη. Άλλο ένα θέμα της έκθεσης είναι ότι γενικώ προχωρούμε καλά οι πολιτικές μας είναι συνεκτικές ό,τι αφορά ε, του στόχου τη της ε, βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά αναρωτιέμαι σε αυτή την έκθεση λαμβάνεται υπόψη τις προσπάθειες που κάνει το Κοινοβούλιο σχετικά. Δηλαδή, έχουμε και εμείς εκθέσεις για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις, ε, τους στόχους. Έχουμε έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων για την κλιματική διπλωματία. Είναι και αυτό ένα κομμάτι των ε, στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε τα θέματα το, της κλωστοφαντουργίας. Είναι πολύ σημαντικά και στην έκθεση αυτή θα βάζατε κάποιες πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου. Έχετε ελέγξει τις εκθέσεις που έχουν υπάρξει συν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί και ο προπολογισμό θα πρέπει να περιλάβει τις, τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχετε χρησιμοποιήσει ως έμπνευση, ας πούμε, ε, τα όσα κάνει το Κοινοβούλιο για να προκύψει τελικώς μια συνεκτικότητα στις πολιτικές μας. Παρόλο βέβαια που το του προσωπικό πλαίσιο δεν είναι μέσω ελέγχου των στόχων, αλλά η δική μας η πολιτική ομάδα, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, έχουν, έχει αναλάβει τέτοιου είδους ε, πρωτοβουλίες ε, για να υπάρξει όντως μια συνέχεια, μια συνεκτικότητα στην ε, πολιτική. Αλλά μπορούμε να μάθουμε ημένα από τους ΔΕ. Οπότε, οπότε ίσω και τα υποδείγματα που μπορεί να αποτελούν κάποιε χώρε αλλά και οι δικέ μα προσπάθειε να μπορούσαν να ενσωματωθούν, να ενταχθούν στην έκθεσή σα. Και τέλο, όταν, μιλούμε, όταν μιλήσαμε στον Φραντ Τίμερμαν, είπε ότι θα ήθελε ε, το θέμα αυτό να το αναλάβει ο οποιοδήποτε αναλάβει μετά από αυτόν. Φαντάζομαι ότι και ο κύριος Βέμπερ είπε κάτι παρόμοιο ε, Ενδιαφέρον λοιπόν θα ήταν, γιατί τώρα μιλούμε για το μετά, αμέσως μετά τις ε, ευρωεκλογέ. Εσείς γνωρίζετε ότι υπάρχουν ε, τέτοιες συζητήσεις ε, στην Κομισιόν για να συμπεριληφθεί στη μετέπειτα δουλειά της το θέμα αυτό και να ασχοληθούν μαζί του οι, τα ύψη στα κλιμάκια της ιεραρχίας και όχι μόνο οι απλοί υπάλληλοι. Εγώ θα ήθελα να συμπεριλάβετε και ε, συναδέλφου εδώ από το ε, Ευρωκοινοβούλιο, τον Κρίστιαν, την ε, ε, αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσει να εμπλουτιστούν. Ευχαριστώ λοιπόν που έχετε προχωρήσει τόσο πολύ όλη αυτή τη διαδικασία. Εγώ ευχαριστώ. Ο Ενρίκη Γκερέρο. Ε, σα ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε να μιλήσω στα ισπανικά, λέει ο μιλητής. Θα μπορούσα ίσως στα γαλλικά, λέει ο μιλητή, αλλά θα προτιμήσω τα ισπανικά. Να ευχαριστήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα για την ενημέρωση, για την ε, δουλειά. Δουλειά η οποία ε, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο μέτρα για να συμμορφωθούμε, αλλά αξιολόγηση για το πού βρισκόμαστε. Και η αξιολόγηση στην ουσία είναι το πρώτο μέτρο που πρέπει να λάβουμε. Γιατί η αξιολόγηση μας λέει ποια είναι η κατάσταση και ποια μέτρα πρέπει να αναλάβουμε ώστε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Και μια καλή αξιολόγηση είναι η πρώτη προϋπόθεση για δέσμευση που έχουμε να λάβει εδώ και 10 χρόνια. Είπατε από την αρχή ότι αυτή η πρώτη αξιολόγηση που θα επαναλαμβάνεται κάθε 4 χρόνια έχει πολλά στοιχεία που άπτονται μια, ε, ενός θετικού παρελθόντος. Και όλα αυτά είναι καλά. Αλλά μετά την παρέμβαση της ΑΝ που γνωρίζει καλύτερα το θέμα, εγώ ήθελα να εκφράσω δύο ανησυχίες, θα έλεγα, θεμελιώδεις. Καταρχάς εγγράφουμε στον κατάλογο των ταπεινών σχετικά με τον άπειρο αυτόν κατάλογο, σχετικά με, τα, με τους στόχους τους βιώσιμους που θέλουμε να επιτύχουμε Καλό είναι που αναλάβουμε αυτές τις δεσμεύσεις, καλό είναι που έχουμε ένα γενικό προσανατολισμό, αλλά εντός 10 ετών σε πολλά μέρη του κόσμου θα είμαστε πάρα πολύ μικρά από τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης. Το άλλο που θέλω να πω είναι σχετικά με το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η δυνατότητα εφαρμογής, υλοποίησης που έχουμε είναι πολύ πιο υψηλή. Και πλησιάζοντας ε, το 2030 Πιστεύω ότι στην πραγματικότητα με την τετραετία αξιολόγηση που θα έχουμε και αντίστοιχα εκείνη που θα έχουμε την οκταετή, θα συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν χώρες που πραγματικά συμμορφώνονται και άλλες που είναι αρκετά μακριά. Θα συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν στόχους που έχουν επιτύχει σχεδόν όλες οι χώρες και άλλοι στόχοι που δεν έχουν πετύχει παρά πάρα πολύ λίγες χώρες. Και επομένως η, ανταπόκριση της κάθε μίας χώρας μεμονωμένα δεν είναι επαρκής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει μια ενουσιακή δέσμευση για να ολοκληρώσει την προσπάθεια των κρατών εκείνων μελών που δεν είναι σε θέση και ο Άρν αναφέρθηκε στην επόμενη Κομισιόν και στην μεταμόρφωση αυτών των στόχων σε μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των 27 ή και 28 που ξέρει κανείς κρατών μελών, ώστε να οικοδομήσουμε το πλαίσιο γύρω από αυτά καθότι δεν έχουμε καταφέρει για τα επόμενα 7 χρόνια άλλη κατεύθυνση να εισαγάμε στο ΠΔΠ, μόνο 3 χρόνια θα έχουμε για να καταβάλουμε μια εντυπωσιακή προσπάθεια, ώστε η χώρα χ που βρίσκεται στην α ή β κατάσταση και που καλείται να καταλαβάλει μια συγκεκριμένη προσπάθεια, να επιτύχει μια εσωτερική αλληλεγγύη και θα το έλεγα καθότι Ισπανός που ζήσαμε τις δεκαετίες του 80 και του 90 τα ταμεία συνοχής ε, ως τεράστια όθηση. Νομίζω λοιπόν θα έχουμε τρία-τέσσερα χρόνια στο τέλος της επόμενης δεκαετίας ώστε να καταβληθεί μια προσπάθεια που, τέτοια που θα βοηθήσει τις χώρες που έχουν καθυστερήσει σχετικά με τους στόχους αυτούς. Ευχαριστώ λέει οι συναλφοί θέτουν μα... μακροσκελή ερωτήματα. Ένα πρακτικό ισοερώτημα. Μιλούμε για τις εξωτερικές πτυχές, αλλά οι εσωτερικές πτυχές πώς θα ενσωματωθούν σε αυτό τον Ιούλιο. Γιατί έχουμε συνάδελφους και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο προσπαθούμε να συμμετάσχουν και άλλοι συνάδελφοι τι ακριβώς Μάλλον καταλαβαίνω ότι θα υπάρχει μια έκθεση για τα εξωτερικά στοιχεία. Για τα εξωτερικά λοιπόν επαναλαμβάνω για τους στόχους του βιωσίμου ανάπτυξης θα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, Να διευκρινίσω καταρχά. Η κοινή σύνοψη αφορά στην εξωτερική πτυχή. Τι θα κάνουμε εξωτερικά για να εφαρμόσουμε το θεματολόγιο. Σημαντικό τμήμα, αλλά μάλλον όχι το πιο δύσκολο. και μάλλον το πιο δύσκολο τμήμα του τεράστιου αυτού θεματολογίου είναι η εσωτερική διάσταση των δεσμεύσεων αυτών. Και σε αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες και στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη. Αλλά είναι μια μακρά διαδικασία, έχουμε πολιτικές σε όλους τους τομείς και πρέπει να τις ενσωματώσουμε και να έχουν μια κεντρική κατεύθυνση. Είχαμε πάρα πολλές σκέψεις για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ανταλλαγή με τον ιδιωτικό τομέα, με διάφορους ενδιαφερομένους κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό το έγγραφο της Κομισιόν που νομίζω ότι πολύ σωστά θέτει τις επιλογές και τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και, λέμε και νομίζω σωστά ότι η επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου θα πρέπει να αποφασίσει πως τα ποια, ποιος ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί. ώστε να αντικατασταθεί, να διαβιβαστεί αν θέλετε πιο κάτω, η στρατηγική 2020. Έχουμε διάφορες επιλογές συνδυασμού, έχουμε σημαντικά ζητήματα πώς θα μεταφράζονται δηλαδή όλα μέσω του θεματολογίου 2030 και εδώ το ζητούμενο είναι πώς μπορούν να ενσωματωθούν αυτά μέσω κεντρικού θεματολογίου ή όχι αλλά αυτή είναι μια συζήτηση την οποία θα πρέπει να διεξιαγάγει η επόμενη Κομισιόν και το επόμενο Κοινοβούλιο. Για να απαντήσω στο τελευταίο σας ερώτημα και ζητώ συγγνώμη που απαντώ κάπως άναρχα αλλά ελπίζω ότι θα τα πω όλα μέχρι το τέλος αν λάβετε υπόψη σας τα δύο παραρτήματα είναι τα όσα είχαμε κάνει στο παρελθόν. Τι κάναμε στόχο προς στόχο δηλαδή. Αυτό θα είναι το περιεχόμενο που θα χρησιμοποιήσουμε για να παρουσιάσουμε τη δράση. Θα υπάρξει επίσης στατιστική ανίσχυση για την νεότερη έκθεση Eurostat που θέλουμε να την έχουμε. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με το Γενικό Γραμματέα για να έχουμε μια κοινή παρουσίαση στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής. με, με, με τρόπο συνεπή και συμπεριληπτικό. Τώρα, για τα εξωτερικά. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι υπερφιλόδοξο. Όλοι αυτοί οι στόχοι για όλες τις χώρες μέχρι το 2030 είναι φιλόδοξο. Το σημαντικό είναι όλες οι χώρες του πλανήτη αυτού να συμφωνήσουν προς ένα όραμα του πού θέλουμε να πάμε. Πρώτα πρέπει να το κάνουμε όλοι αυτό όλοι μαζί. Να την καταβάλουμε αυτή η προσπάθεια και πρέπει να βοηθήσουμε επίσης τις διάφορες τρίτες χώρες να καλύψουν, να επιτύχουν αυτό το θεματολόγιο από μόνες τους. Πρέπει καταρχάς να έχουμε πει και να έχουμε συμφωνήσει ότι αυτό είναι το κοινό θεματολόγιο. Θέλουμε λοιπόν οι δράσει μας οι αναπτυξιακές να είναι ένα μέσο εφαρμογής των στόχων αυτών προκειμένου να επιτύχουμε μία συνένεση. Και μετά αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει αυτό το κοινό θεματολόγιο, αυτό θα πρέπει να διέπει όχι μόνο την διεθνή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την εσωτερική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Και αυτό τώρα πλέον θα πρέπει να αναπτυχθεί, να βρει την αποτύπωσή του σε οποιαδήποτε εθνική πολιτική. Και σωστά τα λέτε, αλλά προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τους στόχους αυτούς στον πραγματισμό, στον διάλογο για τους βιώσιμους στόχους, για τα μετά την Κοτονού, ε, για, τις, ε, για τους μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι χρησιμοποιούμε μια κοινή γλώσσα, κοινό λόγο, προς την κατεύθυνση των αυτών. Πρόκειται για μια συνολική διαδικασία και όταν έλεγα δεν είμαστε ακόμα εκεί, δεν τα έχουμε ακόμα καταφέρει αυτά, εννοούσε ακριβώς αυτό. Έχουμε πολλά στάδια ακόμα μπροστά μας. Τώρα στην κοινή έκθεση προσπαθούμε να αποτυπώσουμε απόψεις του Κοινοβουλίου αναφερόμενοι φυσικά σε μια συνεντική θέση, αλλά θέλουμε να είμαστε και συνοπτικοί. Τι κάνει η Κομισιόν, τι κάνει οι Καρατιμέλη, τι κάνει το Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να είμαστε εξαντλητικοί και υπερπλήρεις. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο αντιπροσωπευτικοί μπορούμε. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι όλα θα αναφέρονται, αλλά μπορώ να υποσχεθώ ότι θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε όλα αυτά που συλλογικώ όλοι από κοινού κάνουμε. Για το επόμενο που πουδουπού, που αυτή τη στιγμή είναι απολύτως υποθετικό, υπάρχει μια πρόταση κομισιόν, δεν υπάρχει καμία απόφαση, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε για πολλά. Ελπίζω να μπορέσουμε στην επόμενη θητεία στην επόμενη έκθεση μάλλον να πούμε περισσότερα για το πι γιατί σε αυτήν εδώ δεν μπορούμε. Αυτά από πλευρά Ωραία. Θα, είναι, θα έχουμε δύο σημαντικές λοιπόν συναντήσεις το καλοκαίρι. Και το Κοινοβούλιο βεβαίως θα εμπλακεί. Και ελπίζω ότι θα εμπλακούν και άλλες περισσότερες ε, επιτροπές γιατί είναι σημαντική η δουλειά. Ευχαριστώ και τους δύο, την ομάδα της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Ελπίζουμε ότι οι καρποί των ε, προσπαθειών μας θα έρθουν σύντομα όπως είπε και ο και είναι πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει αλλά είναι ο μόνος τρόπος αυτός. Ακόμα και παρά τις επιθέσεις στην πολυμέρεια που βλέπουμε καθημερινά η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαριστούμε λοιπόν και την Κομισιόν και την ΕΕΔ. Στι 6.30 έχουμε μία δεξίωση. Η Κομισιόν ε, είσαστε προσκεκλημένοι. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Προχωρούμε. Βλέπω πολλούς προσκεκλημένους σήμερα από την κοινότητα των Γεζίντι. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Πριν έρθουμε στο δικό σας σημείο, κάντε λίγο υπομονή σας παρακαλώ. Πάμε στο σημείο 7 για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Νότιο Αφρική, Μαλάουι, Μοζαμβίκη και Ζιμπάμπουε μετά τον κυκλώνα. Θα είδατε φαντάζομαι πολύ με τρόμο στις τηλεοράσεις τις εικόνες που χτύπησαν από τον κυκλώνα, ο οποίος κατέστρεψε μεγάλα σημεία. Χτύπησε την ε, περιοχή της Μπέιρα, στην κεντρική Μοζαμβίκη. Ε, κατέστρεψε χωριά δίπλα στις περιοχές Σοφάλα, Μανίκα, Ζαμπίζια, Τέτε και Ινχαμπάνε. Επλήγησαν από ε, πλημμύρες. Δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα επίσης και στην Μανικαλάνδη και το Μασφίγγο. Μέχρι στιγμής τα θύματα έχουν φτάσει τους 446 ανθρώπους στη Μοζαμβίκη και 154 στη Ζιμπάμπουε. Είναι πραγματικά η χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή που σχετίζεται με τον, καιρό, με τον στο νότιο ημισφαίριο. Βεβαίως, ε, προς το παρόν, ε, όλοι έχουν στο κέντρο των προσπαθειών την ε, ανθρωπιστική ανταπόκριση. Αλλά βεβαίω είναι και μακροπρόθεσμο το έργο που πρέπει να γίνει ε, γιατί χάσει, έχουν χάσει οι άνθρωποι το βιό του, τις ε, ε, φυτίες τους, τα ζώα τους και ξέρουμε ότι ούτω ή άλλω κάποιε από αυτέ τις χώρες είχαν ήδη προβλήματα να αντιμετωπίζουν με ασθένειες κλπ. Οπότε... Εγώ ε, έχω έρθει σε επαφή με τον Επίτροπο Στυλιανίδη και εντό λίγων ωρών μετά την καταστροφή ε, απάντησε και έστειλε τις, ε, δωμά, τις μονάδες. Τώρα έχουμε την Ντομινίκ Αλμπέρ εδώ, ε, επικεφαλής της μονάδας για την Ανατολική και Νότιο Αφρική, της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ, για να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς, αλλά και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτή την καταστροφή. Έχετε το λόγο κυρία Αλμπέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια σύντομη ενημέρωση για το πώς έχει η κατάσταση τώρα θα σας κάνω, θα σας πω τι έχει γίνει από πλευράς ανταπόκρισης μέχρι στιγμής και θα σας πω τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος. Αυτό που βλέπετε στις ε, διαφάνειες είναι από τις φωτογραφίες από τους εμπειρογνώμονες ε, ε, της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ λίγες ώρες μετά την, τον κυκλώνα στην Μπέιρα, στη Μοζαμβίκη. Έτσι ήταν η κατάσταση εκεί, όπως τη βλέπετε στη διαφάνεια. Δεν μιλούμε μόνο για τη Μοζαμβίκη βέβαια, μιλούμε και για το Μαλάουι και για τη Ζιμπάμπουε. Ο τροπικός κυκλώνας Ιντάι χτύπησε την 14η ε, Μαρτίου την ε, πόλη της Μπέιρα στη Μοζαμβίκη με καταστροφικές βροχές ε, και ανέμους. Συνέχισε προς τα ανατολικά και έφτασε στη Ζιμπάμπουε. Από τις αρχές Μαρτίου έχουν υπάρξει σημαντικέ ε, βροχοπτώσει ε, στο Μαλάουι και τη Μοζαμβίκη που από κοινού με τον ε, κυκλώνα δημιούργησαν τεράστιες πλημμύρες στις δύο αυτές χώρες. Ο αντίκτυπο λοιπόν είναι, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο όσο έρχονται όλο και περισσότερε πληροφορίε από την περιοχή. Η κατάσταση σήμερα στη Μοζαμβίκη δείχνει ότι έχουν υπάρξει πάνω από 500 θύματα, πάνω από 794.000 επλήγησαν από τις πλημμύρες και από τον κυκλώνα. 141.000 άνθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια, ε, έχει μπει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Μοζαμβίκη και οι περισσότεροι από αυτούς που επλήγησαν από τον κυκλώνα ε, είναι γεωργοί, έχουν πάνω από 500.000 εκτάρια καταστραφή λόγω του κυκλώνα και έχουμε πρόβλημα με τους ανθρώπους γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό στην Μπέιρα αλλά και σε άλλες περιοχές. Η Μπέιρα ε, πραγματικά ε, πλήγει σημαντικά, όπως βλέπετε και στην, όπως είδατε μάλλον στην φωτογραφία πιο πριν. Η ε, αναδόμηση των κρίσιμων υποδομών όμως έγινε πολύ γρήγορα Τώρα με τις υπηρεσίες ε, των σιδηροδρομικών σταθμών ε, λειτουργούν ε, ο και τα, και, το αεροπλα... και τα αεροδρόμια επίσης είναι 100% λειτουργικά. Στο Μαλάουι οι πλημμύρες δημιούργησαν εκτοπισμό. Πάνω από 86.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν από τις αστείες τους και 800.000 άνθρωποι επλήγησαν συνολικά. Και πάλι η κυβέρνηση έθεσε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κατάσταση σιγά σιγά επιτόπου βελτιώνεται. Όλες οι πληγήσει περιοχέ ε, στις ανατολικά του ποταμού που ήταν προσβάσιμες μόνο μέσω α, α, σκαφών μέχρι τι 21 ε, Μαρτίου τώρα α, μπορούν και να ε, είναι προσβάσιμες και οδικώ. Στην Ζιμπάμπουε έχουμε 320 ανθρώπους που είναι αγνοούμενοι, 270.000 άτομα έχουν πληγεί και ο πρόεδρος της Ζιμπάμπουε πάλι έχει θέσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η αξιολόγηση βεβαίω τη κατάσταση ε, συνεχίζεται στη Ζιμπάμπουε. Η πρόσβαση είναι πραγματικά το πιο σημαντικό πρόβλημα που καθιστά βεβαίω και την ε, κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Ε, είναι σημαντικέ οι ζημίε στι υποδομέ και ο κυκλώνα χτύπησε μια περιοχή που είχε ούτω ή άλλω πληγεί από θέματα, για, λόγω προβλημάτων ασφάλειας αλλά και α, διατροφικής ασφάλειας. Τώρα, η άμεση απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ ανέπτυξε διάφορους ε, εμπειρογνώμονες ε, και τον ε, αξιωματούχο επικοινωνίας στις τρεις χώρες για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα της κατάστασης επιτόπου. Το, η υπηρεσία Κοπέρνικους κινητοποιήθηκε. Είναι η υπηρεσία που παράγει χάρτες. Οπότε δημιουργήθηκαν πάνω από 50 χάρτες για τις περιοχές και πραγματικά απεδείχθησαν πάρα πολύ χρήσιμοι για τις ε, κυβερνήσεις των τριών αυτών χωρών για να μπορέσουν να σχεδιάσουν και να υποστηρίξουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποίησε και επιπλέον χρηματοδότηση για να αντιμετωπίσει την, ε, τις έκτακτες αυτές ανάγκες. 3,5 εκατομμύρια ευρώ, 2 εκατομμύρια πήγαν στη Μοζαμβίκη, ένα στο Μαλαούι και μισό στη μισό εκατομμύριο στη Ζιμπάμπουε. Στη Ζιμπάμπουε. Ε, επικεντρωθήκαμε λοιπόν στα θέματα επιμελητία που ήταν βασική ανάγκη στην αρχή, αλλά βεβαίω και σε πολυτομεακή στήριξη. Επιπλέον βεβαίω τη ε, στήριξη του IFFC, του Ερυθρού Σταυρού στη Μαλάουι και τη Μοζαμβίκη, που ήταν ούτω ή άλλω από την αρχή πολύ ενεργοί στην ανταπόκρισή του. Εδώ βλέπετε τα ελικόπτερα της ΕΚΟ που ε, παραδίνουν, παραδίνουν τη βοήθεια στην Ζιμπάμπουε σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες ακριβώς μετά την ε, έλευση του κυκλώνα. Εδώ βλέπετε το, ε, ε, το σύστημα εξυγένσης υδάτων, το οποίο δημιουργήθηκε και παραδόθηκε μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Και με την έκτατη αυτή χρηματοδότηση στηρίζουμε και τον Ισπανικό Ερυθρό Σταυρό στη Μοζαμβίκη, που συνεργάζεται στενά με τον Ερυθρό Σταυρό με, της Μοζαμβίκης για να υπάρξει πρόσβαση σε άτομα όπου υπάρχουν, σε, σε περιοχές όπου υπάρχουν εκτοπισμένοι. Και μπορεί να το ξέρετε ότι ήδη υπάρχουν κρούσματα χολέρας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να το προωθήσουμε αυτό. Και επίσης σημαντικό είναι να ξέρετε ότι ε, όσοι έχουν εγκατασταθεί στα σχολεία θα θέλαμε να ε, επανέλθουν στις αιστείες τους, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και πάλι τα σχολεία. Αλλά δυστυχώς οι εκτοπισμένοι έχουν χάσει τα πάντα. Εδώ βλέπετε τα εγγένεια της ε, λειτουργίας της μονάδας των, της Ιταλικής για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ε, βλέπετε την συνέντευξη που δόθηκε. Εδώ βλέπετε τη χρήση drone και εξοπλισμό, εξοπλισμό από τον WFP, από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων, για να αξιολογηθεί η ζημιά και η κατάσταση στις ε, περιοχές για να δούνε αν μπορούν οι εκτοπισμένοι να επιστρέψουν στις αιστείε τους, αν είναι προσβάσιμε οι σε περιοχές οδικός ή όχι. Εδώ βλέπετε ε, Η πορτογαλική ομάδα είναι αυτή που βλέπετε, με πυροσβέστες που ε, καθαρίζουν τα πεσμένα δέντρα και τις ζημιές ε, τις πρώτες, ε, την πρώτη εβδομάδα μετά την, τις έκτακτες αυτές συνθήκες. Έφυγαν τώρα από την Πέιρα, αλλά έχουν αντικατασταθεί από μια ομάδα έκτακτη που ασχολείται με την παροχή ιατρικής βοήθειας. Τώρα, για την άμεση ανταπόκριση, το ενδιαφέρον είναι το εξή. Από τη μια υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια, από την άλλη Υπάρχει πολιτική προστασία και η ανταπόκριση της Ευρωπαϊ... του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε από την κυβέρνηση της Μοζαμβίκης άμεσα. Η βοήθεια δόθηκε μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και περιλαμβάνει διάφορες δυνατότητες, ε, ε, συστήματα εξυγένσης νερού, νοσοκομιακή βοήθεια, έκτακτες ιατρικές μονάδες τηλεπικοινωνίες, ε, δουλειά πάνω στις τηλεπικοινωνίες και στην αποκατάσταση του ίντερνετ. Εννέα κρατημέλη παρέχουν βοήθεια μέσω του, πολιτισμού, του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Και η Επιτροπή επίσης ε, έστειλε και μία πλήρη ομάδα μελή, για να συντονίσει την, ε, την ανταπόκριση και να βοηθήσει την κυβέρνηση της Μοζαμβίκης. Η ανταπόκριση βεβαίω δεν έχει ολοκληρώσει. Ε, πρέπει να αξιολογηθεί φυσικά το τι έχει γίνει. Να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες ε, που έχουν παραμείνει. Είναι τα αντικουνουπικά, γιατί η ελονοσία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ε, υγειονομικά κιτ, σετ για την κουζίνα ε, βοήθεια προς τα, για, την, ε, για τρόφιμα. Επίσης, ε, μια ομάδα μας αναφέρει ότι σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες εξυγίανσης είναι τα πράγματα εντάξει πια. Και αυτό κατέστη δυνατό ακριβώς λόγω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης που έστειλε τον εξοπλισμό. Επίσης, για τους εκτοπισμένους πρέπει να δούμε θέματα προστασίας τους. Έχουν ε, εκτοπιστεί, προς το παρόν μένουν σε κάποια ως προσωρινούς καταβλισμούς και βεβαίως ο, κίνη, ο κίνδυνος σεξουαλικής βίας και βίας ε, με, το φύλλο είναι πολύ μεγάλος. Ε, παιδιά μικρά έχουν χαθεί από τους γονείς τους, ηλικιωμένοι επίσης είναι έχουν σημαντικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Οπότε πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προκλήσεις. Χολέρα. Κρούσματα χολέρας έχουν παρατηρηθεί στην Πέιρα, αλλά μπορεί να μην είναι μόνο στην Πέιρα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις διάρειας, ελονοσία επίσης, κρούσματα ελονοσίας που μας ανησυχούν. Στη Ζιμπάμπουε ο κυκλώνας συνέβη μετά από μια δύσκολη κατάσταση στη χώρα για, το, για θέματα ε, υποσυντισμού, ασφάλειας τροφίμων, επιστηστικής ασφάλειας και έτσι η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. Δεν πρόκειται να βελτιωθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες γιατί έχουν καταστραφεί οι εισοδιές λόγω των πλημμυρών και επίσης γιατί ε, ετοιμάζονταν να ε, ε, συλλέξουν τις σοδιές, οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Επίσης η εκπαίδευση έχει σταματήσει. Τα σχολεία πια χρησιμοποιούνται ως κέντρα εκένωσης. Πρέπει να αρχίσουν να ξαναλειτουργούν και πάλι ως σχολεία. Και συνολικά ακόμη και παρά το γεγονός ε, ότι ξέρουμε ότι περνάει γρήγορο καιρό, τα πράγματα ε, ακόμη εξελίσσονται. Εμείς συνεχίζουμε να αναλύουμε την κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται και όσο παίρνουμε περισσότερες πληροφορίες από τις επιτόπου ομάδες. Τώρα, για τα επόμενα βήματα. Για μας, τι θα πει αυτό. Θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των ομάδων πολιτική προστασία. Έχουμε κάποιε μονάδε οι οποίε θα αποσταλούν στι χώρε. Για τα ανθρωπιστικά θέματα θα συνεχιστεί βεβαίω και η προσπάθεια ε, για να, πάρουμε, για να έχουμε υπόψη μα και την ανταπόκριση για την αντιμετώπιση τη ε, χολέρας και πιο μεσοπρόθεσμα ή και πιο μακροπρόθεσμα ε, αν, ε, αντιμετώπιση ε, επανα επανεγκατάσταση των ανθρώπων στις αιστείες τους, ε, προγράμματα αντιμετώπισης ε, ε, κλιματικών καταστροφών και δημιουργίας αντίστασης σε τέτοιου είδους καταστροφές, γιατί μια φυσική καταστροφή θα ξανασυμβεί. Αυτά συνολικά από μένα, έτσι μια γενική εικόνα, Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πλήρες η ανάλυση που μας κάνατε. Είδαμε και τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Ο Ενρίκη Γκερέρο είναι ο εισηγητής, οπότε να του δώσουμε το λόγο. Σε eh, Ευχαριστώ για τις ε, πληροφορίες αυτές. Θα ήθελα να πω ότι νιώθω μια δυσφορία. Νομίζω όλοι τι νιώθουμε όταν βλέπουμε να συμβαίνουν τέτοιου είδους καταστροφές και πώς αυτές οι τεράστιες καταστροφές δημιουργούν τελικά ελάχιστο, προκαλούν ελάχιστο ενδιαφέρον στις χώρες μας. Όταν γίνεται μια τρομοκρατική επίθεση σε οποιαδήποτε χώρα, στην Ισπανία ας πούμε, Μπορεί να έχουμε νεκρού. τέσσερι ανθρώπου, ας πούμε, που είναι βεβαίω τραγικό, αλλά γίνεται παγκόσμια είδηση. Γίνεται είδηση τουλάχιστον σίγουρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν πεθαίνουν χιλιάδε επειδή έχει χτυπήσει ένας τυφώνας μια χώρα, το παίρνουμε σαν να ήταν απλώς μια φυσική καταστροφή, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, δεν μπορούμε να τις αποτρέψουμε τέτοιου είδους καταστροφές στο μέλλον, οπότε δεν ασχολούμαστε. Ένα από τα αριθμητικά στοιχεία που μας είπατε δείχνουν ότι στο Μαλάουι μόνο υπάρχουν άνθρωποι που ε, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που, είναι, που έχουν πληγεί, που είναι ε, ίσοι με, τους, με όσους όλους τους πρόσφυγες που έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν σε μια χώρα μέσα σε τρεις ημέρες ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν πληγεί είναι τόσο μεγάλος και ίσως ουσιαστικά με τους πρόσφυγες που έχουν φτάσει στα σύνορα της Ευρώπης. Ε, όταν βλέπουμε τέτοιου είδους ε, κρίσεις, τέτοιου είδους καταστροφές, καταλαβαίνουμε πόσο επιδεινώνεται η κατάσταση σε, μια, σε κάποιες χώρες που ούτως ή άλλως ήταν δύσκολη. Ε, ή από την ε, ανθρωπιστική πλευρά ή από την πλευρά της ιατρικής περίθαλψης. Υπάρχει καταστροφή στον τομέα της παιδείας. Ούτως ή άλλως ο πληθυσμός είχε προβλήματα πρόσβασης στην ε, εκπαίδευση. Ή στέγαση επίσης. Η καταστροφή, η ζημία στην γεωργία σε χώρες που πριν από το χτύπημα του κυκλώνα είχαν σημαντικές δυσκολίες να ε, παράσχουν τρόφιμα σε όλους τους πολίτες τους. Το μόνο καλό νέο είναι ότι σε κάθε χώρα έχουν υπάρξει ενδείξεις αλληλεγγύης, ανεπαρκείς μεν σε ποιοτικό επίπεδο, αλλά παρόλα αυτά είναι καλό να βλέπουμε τέτοια δείγματα ότι όντω υπάρχει αλληλεγγύη. Είδαμε την Ιταλική ομάδα να δίνει βοήθεια, τον Ισπανικό Ερυθρό Σταυρό να συμμετέχει, ομάδες ε, ιατρικές από την Πορτογαλία. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε θετικά. Αλλά δεδομένου και του όγκου της καταστροφής, τα κονδύλια που έχουμε καταφέρει να κινητοποιήσουμε είναι σταγόνα στον ωκεανό. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε σχέση με το τι μπορούμε να καλύψουμε με αυτά τα κονδύλια. Αν λοιπόν ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο ιατρικής περίθαλψης, ή αγροτικής παραγωγής, αν προσπαθούμε να παράσχουμε στο ένα ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευση σε αυτέ τι τάξει των σχολείων που έχουν καταστραφεί, θα πρέπει όντω να, να, να εντείνουμε τι προσπάθειε επανένταξη τώρα. Το θέμα δεν είναι απλώ να ανταποκριθούμε στην έλλειψη νερού ή να αντιμετωπίσουμε τα κρούσματα χολέρα. Βεβαίω είναι και αυτά επίγοντα, αλλά αντιμετωπίσουμε τεράστιου μεγέθους κρίση. Και αυτό θα επηρεάσει και εμάς και τις ίδιες τις χώρες για πολλά χρόνια. Και θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα της στρατηγικής μας για τη μελλοντική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αυτών, και τη συνεργασία τους με αυτές τις χώρες. Έχω, νομίζω, λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Θα είναι μάλλον η τελευταία μου παρέμβαση στο Κοινοβούλιο. Είμαι εδώ 10 χρόνια. Πάντα ήμουν μέλος της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Στην αρχή ήμουνα ε, παρατηρητής, ήμουνα επισκέπτης στην ΑΦΚΟ τα πρώτα χρόνια, ήμουνα μέλος της ε, Επιτροπής ΔΕΒΕ. Έχω συνεισφέρει με τη βοήθεια όλων βεβαίως, έτσι ώστε κάτι να μπορέσουμε να κάνουμε για τις διάφορες καταστροφές που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Ήμουν εισηγητή για την ανθρωπιστική βοήθεια και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη τη Επιτροπή μα. Πραγματικά πάντα ήταν διατεθειμένα να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Όπω ο Ενρίκε που ασχολείται με τα θέματα τη ανθρωπιστική βοήθεια, όχι επειδή δεν τον αναφέρω επειδή είναι Ισπανό συμπατριώτη, αλλά ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί ήταν σημαντική η βοήθειά του, αλλά και όλα βεβαίω τα μέλη τη Επιτροπή ΝΤΕΒΕ. Πάντα λέγαμε ότι αυτή η Επιτροπή είναι πολύ ιδιαίτερη Επιτροπή οι ιδεολογικές ε, διαφορές και οι ε, οποιοδήποτε άλλου είδους διαφορές μπαίνουν στην άκρη και μπορούμε εδώ να συνεργαστούμε παρά τα όσα μας χωρίζουν. Και επίσης να ευχαριστήσω και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Έχω συνεργαστεί με κάποιους από εσάς, ειδικά με το Ρενό που είναι και εδώ σήμερα. Εγώ δεν θα είμαι εδώ στο μέλλον, αλλά θα προσπαθώ να βοηθώ όπως μπορώ για όλα αυτά τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε σε αυτή την Επιτροπή. Ενδίκε, ήμουν έτοιμη να πω, μας είχες πει ότι πρέπει να φύγεις 4.30 γιατί έχεις άλλη ανηλυμένη, αλλά θα μας λείψεις. Εγώ δεν θα είμαι εδώ λέει η πρόεδρος, αλλά όλοι μου λένε και ε, τα μέλη του προσωπικού της γραμματείας ότι θα μας λείψει ο Ενρίκε. Γιατί έχεις όλα αυτά τα μεγίστα δάχτυλά σου. Για τη Μοζαμβίκη, τα υπόλοιπα. Και όλα αυτά, όλοι αυτοί οι αριθμοί σημαίνουν ανθρώπους, πραγματικές οικογένειες, ζωές που χρειάζονται τη βοήθειά μας. και νομίζω ότι πάντα καταφέρνεις να βρίσκεις έναν τρόπο να καταδεικνύεις πράγματα που είναι πραγματικά πολιτικά ζητήματα και που πρέπει πραγματικά να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι σε όλα αυτά τα ανθρωπιστικά ζητήματα, τα ζητήματα πραγματικής ανάπτυξης πάντα έδειξε... το ανθρώπινο πρόσωπο του Κοινοβουλίου. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε και στα πρακτικά Εξαιρετικό συνάδελφος ο Ενρίκε. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Δεν θα είναι εδώ απόψε και άρα έπρεπε να τον ευχαριστήσω τώρα. Τζούντεθ Αργεντίνη τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση των έκτων μέτρων που έλαβε η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Θυμάμαι το 2000, όταν μόλις ξεκινούσα, σε μια μη μικρων ε, αναπτυξιακής βοήθειας, ε, τεράστια προβλήματα για τη Μοζαμβίκη. 19 χρόνια αργότερα, αντίστοιχα πράγματα βλέπουμε. Μήπως πρέπει να πούμε δύο λόγια και για την ετοιμότητα και για την κλιματική αλλαγή. Γιατί όλα αυτά ανά 20 χρόνια σημαίνουν εξαιρετικά μεγάλη πρόκληση για μια χώρα. Και υπάρχει μια κατανόηση για την επόμενη μέρα. Υπάρχει μια επίγουσα ανάγκη για την οποία και ευχαριστούμε. Αλλά τι σημαίνουν αυτά για την περαιτέρω ανάπτυξη στην όλη περιοχή. Νομίζω ότι θα έχουν βουλευτικές εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αν δεν απατώμα. Αλλά όλα αυτά μάλλον σημαίνουν σημαντικό πισωγύρισμα για την κανονική λειτουργία της χώρας αυτής. Κάνατε και την ε, διασύνδεση με τη Ζιμπάμπουε, με τις ταραχές λόγω των υψηλωτάτων τιμών των καυσίμων και πέραν αυτού. Δεν ξέρω αν βλέπετε και άλλες ομοιότητες με την ε, Μοζαμβίκη. Και τι γίνεται και με το Μαλαουί γιατί αυτή είναι μια άλλη χώρα που πρέπει να έχει επηρεαστεί έντονα από αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και στην Τζούντιθ πάνε οι ευχαριστίες μας, προφανώς. Αυτά συνήθως τα θυμόμαστε στις τελευταίες συνεδριάσεις, στις τελευταίες συναντήσεις, αλλά είχατε κάνει και για τα ορυκτά πολύ σημαντικά πράγματα, πολύ σημαντική δουλειά για την ευθύνη που έχουμε, να πηγαίνουν οι αναπτυξιακοί πόροι, η αναπτυξιακή ενίσχυση εκεί που πρέπει. Τζούντιθ Argentini λοιπόν, 10 χρόνια είναι μαζί μας, αν δεν κάνω λάθος, και επίσης θα αποχωρήσει. Ένα από τα νέα μέλη τώρα, η Μέλια Μπέκα πέρα, ευχαριστώ πρόεδρε, λέει η κυρία Μπέκα πέρα, αυτή η καταστροφή ε, μεταξύ, μάλλον στην ε, Νότια Αφρική, στην περιοχή της Νότια ε, μας σοκάρει όλους και νομίζω ότι πρέπει να αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο στην πολιτική μας δουλειά, στο πολιτικό μας έργο. Πρόκειται για μια πραγματικά μεγάλη έκταση καταστροφή με χίλια θύματα το οποίο είναι πραγματικά τραγικό. Οι πόροι λοιπόν ρωτώ που αποστέλουμε τι όλη βοήθεια, η όλη ενίσχυση είναι επαρκής. Μήπως θα έπρεπε να είναι πιο μεγάλη. Θα ήταν δυνατόν να αυξήσουμε την ενίσχυσή μας. Επίσης η ανοικοδόμηση που είναι μια τεράστια προσπάθεια πόσα χρόνια θα χρειαστεί να εργαστούμε στην προσπάθεια της ανοικοδόμησης και τι διαστάσεις είναι αυτής η προσπάθειας. Τι, τι, για τι είδους πόρους μιλούμε. Σας ευχαριστώ. Ανιλίτς επίσης βεβαίως. Πρόεδρε, με μία φράση θα υπογράμμιζα την πολύ μεγάλη δουλειά του Ενίκε και της κυρίας ε, Σαρτζεντίνη μέσω των οποίων γνωρίσαμε και πολλά καινούργια μέλη στη δουλειά αυτή. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, πολυπίκυλη αυτή δουλειά και προσπάθεια που έχετε κάνει. Οι τελευταίες ερωτήσεις με βρίσκουν σύμφωνο, δεν θα τις επαναλάβω. Και για μένα είναι θέμα περισσότερο διαμόρφωση πολιτικής. Από την ΕΝΒΙ και από την ΑΦΕΤ χρησιμοποιούμε περισσότερο την διπλωματική οδό την οποία ακολούθησε και η Σουηδία και η Γερμανία, που συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Έθνη για να βελτιώσουν τον μικρομηχανισμό της κλιματικής αλλαγής και τι πρέπει να αλλάξουμε ώστε να αποτρέψουμε περιπλοκές που προκύπτουν από τέτοιου είδους επεισόδια κρούσματα. Είχαμε συμπεράσματα του Συμβουλίου για το κλίμα και ιδιαίτερα για την πολιτική για το νερό. Ιδιαίτερα. Πιο ειδικά δηλαδή. Επί του οποίου ρωτώ και την ΙΕΔ και την Κομισιόν. Πιστεύετε ότι εφαρμόζοντας αυτό το σκεπτικό για την μεγαλύτερη διπλωματική συνέπεια πρέπει να έχουμε για την κλιματική αλλαγή και για το πώς εφαρμόζουμε τις ενισχύσεις που δίνουμε σε χώρες για το αυξημένο δυναμικό απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα έχουμε την υποστήριξη των κρατών μελών. Έχετε συζητήσει για την συνέπεια του φάσματος πολιτικής, για την ανάπτυξη του δυναμικού, όχι μόνο αυτά δηλαδή που συζητά η Σουηδία και η Γερμανία με το Ηνωμένα Έθνη, αλλά και πέραν αυτού εξετάζοντας την κατάσταση της Μοζαμβίκης μήπως θα, έχουμε, μήπως θα έπρεπε να είχαμε μια προσέγγιση περισσότερο εδρασμένη, βασισμένη στην γνώση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Αλμπέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα σχολιάσω τα των δημοσιευμάτων του τύπου, αλλά τα της αλληλεγγύης, γιατί ήταν κάτι που ήταν άμεσα προφανές στην ανταπόκριση προς την κρίση αυτή. Το γεγονός ότι έχουμε εννέα κράτη-μέλη που κινητοποίησαν τις ομάδες πολιτικής προστασίας ε, για να συντονιστούν ήταν κάτι απτό και προφανές από τους ίδιους κατοίκους της χώρας. Ως απτή αλληλεγγύη, απτή βοήθεια που προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρομαι. Τώρα, για μέσο μακροπρόθεσμες ε, προοπτικές, να πω ότι πράγματι η περιφέρεια της Αφρικής και οι δύο ειδικά χώρες αυτές είναι εξαιρετικά εκτεθειμένες στον κίνδυνο Πράγματι έχουμε τώρα μια εξαιρετική περίπτωση κρούσματος, αλλά είχε συμβεί στο παρελθόν, θα συμβεί στο μέλλον. Υπό την οπτική της ΓΔΕΚΟ το εξετάζουμε με τα μέσα που έχουμε διάθεσή μας, δηλαδή κυρίως εργαζόμαστε στα θέματα ετοιμότητος αντιμετώπισης κρίσεων. Αυτό κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Επομένως, η εστίαση, η προσοχή είναι στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του, της ε, εθνικής δυνατότητας να ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές. Αυτό δεν το κάνουμε με μονομένα απομονωμένα, μαζί με τις κυβερνητικές αρχές και μαζί με τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες. γιατί αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο συντονισμένα μέσω μιας συνολικής ανθρωποστικής προσπάθειας. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε επαναλαμβανόμενες κρίσεις είναι στο κέντρο αυτής της προσέγγισης που έχουμε αναπτύξει. Για την συνέπεια της πολιτικής φοβούμε ότι αυτό περισσότερο θα ενέπιπτε στην αρμοδιότητα των συναλήφων της ΙΕΔ ή της ΔΕΒΚΟ που ίσως δεν είναι εδώ, αλλά εγώ μπορώ να μιλήσω για τα θέματα ετοιμότητος. Για τα διατροφικά, όσο γάμα δελτα ίσως να ξέρετε ότι έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό συνεργατών Ε, σχετικά με τη δυνατότητα που έχουν να ανταποκρίνονται όταν εμφανίζεται το πρόβλημα. Είναι κάτι δηλαδή επί του οποίου έχουμε υψηλή ευαισθητοποίηση, έχουμε λάβει κάποια μέτρα μετά το κρούσμα αυτό και ναι, προσπαθούμε μέσω των εταίρων που χρηματοδοτούμε αυτή τη στιγμή να το λάβουμε αυτό υπόψη μας και να μην ξαναπέσουμε αν θέλετε στις ιστερήσεις του παρελθόντος. Κατά πόσον η ενίσχυση που παρέχουμε αυτή τη στιγμή είναι επαρκής, σίγουρα όχι. Αλλά η Κομισιόν δεν είναι μόνη της. Κάτι που κάνουμε από την αρχή της κρίσης είναι να υποστηρίζουμε και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να έχουμε μια πληρέστερη ενίσχυση, ανταπόκριση. Αυτό θα συνεχιστεί. Και θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ενίσχυση αυτή συνολικά. Η ανοικοδόμηση πράγματι είναι μια σημαντική πρόκληση. Αυτό θα αντιμετωπίσουμε στους επόμενους κύκλους μαζί με τους συναδέλφους της ανάπτυξης. Οι συνάδελφοι της Devco από την αρχή συνεργάζονται μαζί μας, από την αρχή της κρίσης, γιατί είναι σημαντικό να έχουν λάβει υπόψη τους την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προκειμένου να αναπτύξουν οποιαδήποτε αναπτυξιακά προγράμματα. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε πόσο αποτελεσματική είναι η ΕΚΟ στον συντονισμό να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μας και στους συνεδέλφους σας στο πεδίο γιατί ξέρουμε ότι πολύ συχνά είναι δύσκολες συνθήκες, καλούνται να κάνουν δύσκολα πράγματα. Ευχαριστούμε λοιπόν και με αυτό συνάδελφοι ολοκληρώσαμε με το, με το σημείο 7 και μπορούμε να πάμε στο σημείο 8. Περιμένω απλώς ένα λεπτό τους προσκεκλημένους στο πανέλ γιατί ξέρω ότι υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον. Okay, um, thank Θα προχωρήσουμε τώρα να συζητήσουμε για ένα άλλο δύσκολο ανθρωπιστικό θέμα, το υπαριθμόν 8, για την κατάσταση των Γιασίδη στο Ιράκ. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το λόγιο στους μας, τα, την κουρδική μετάφραση είναι το κανάλι 25. Μπορείτε να παρακολουθήσετε λοιπόν μετάφραση στην κουρδική γλώσσα στο, ε, στο κανάλι 25. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την κουρδική μετάφραση. 25 λοιπόν. Και για να μιλήσετε Άρα, ναι, θα μεταφράσετε και τις άλλες γλώσσες από τα κουρδικά. Ωραία. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στη συζήτηση που ε, ε, ε, έγκυται σε ανταλλαγή απόψεων με το Κεντρικό Συμβούλιο των Γεζίντι στην Γερμανία, που είναι το όργανο που εκπροσωπεί τους Γεζίντι, τις κοινότητες Γεζίντι στο Ιράκ και αλλού. Καλωσορίζω λοιπόν τον Δόκτρα Ιρφάν Οτάκ, επικεφαλής του Συμβουλίου και τον κύριο Μαρουάν Σάμπρι Μπαντάλ, καλώς ήρθατε, που είναι διακεκριμένος ηγέτης της κοινότητας Γιασίδη στο βόρειο Ιράκ, η οποία κοινότητα υπέστη επίθεση από το Ισλαμικό κράτος το 2014 με αποτέλεσμα πολλούς θανάτους Γιασίδη. Μετά οργανώθηκε αντίσταση κατά του Ισλαμικού κράτους. και μπόρεσαν να απελευθερώσουν και πολλές κρατούμενες γυναίκες για σύντη με ε, τον κύριο Μαρουάν που ε, υποδεχθήκαν προηγουμένω. Είμαι βέβαια ότι καλύτερα θα μπορέσετε να τα εξηγήσετε εσεί ε, τα, τον Γιασίδη. Εισαγωγικά, η Γιασίδη είναι περίπου ένα εκατομμύριο ψυχέ στο, στον κόσμο όλο, 750.000 στο βορειοδυτικό Ιράκ, άλλε κοινότητε βρίσκονται στη Συρία, Τουρκία και Ιράν και πρόκειται για ε, θρησκευτική μειονότητα και πολλοί ζουν τώρα και στο εξωτερικό και ιδίως στην Γερμανία. Υπάρχουν επίσης κοινότητες στην Αρμενία, Γεωργία και Ρωσία αλλά και σε άλλες χώρες της Αιγής Ανατολής. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κατέστη γνωστή η δυσμενής μοίρα ε, των Γιασίδη στην κρίση στην Αιγής Ανατολή όταν ήλθε η Νάντια Μουράτ για να τη απονεμηθεί το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία σκέψη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα λησμονήσω ποτέ ε, που άκουσα την ιστορία της Νάντια Μουράτ όταν ε, το πρόσωπο αυτό μίλησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει λάβει τώρα ε, το Δαμακουίγκι το βραβείο Νομπέλ. Είχε πει ότι ήθελε να πει τι έγινε, αλλά ήθελε και δικαιοσύνη για τον λαό τη. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ικανοποιημένη που θα διεξαχθεί η συζήτηση αυτή σήμερα και θα μπορέσουμε να ακούσουμε για την τρέχουσα κατάσταση των Γιασίδη στο Ιράκ. Περίπου 400.000 άνθρωποι εκτοπισμένοι σε καταβλισμούς προσφύγων σε ολόκληρο το Ιράκ και σε ορισμένα τμήματα του Κουρδιστάν. Ε, χαίρομαι λοιπόν που είστε παρούσες και παρόντες εδώ και ελπίζω θα μπορέσουμε να ακούσουμε και θα μπορέσουμε να ακούσουμε από τον κύριο Σάμπρι Βαντάλ θα είναι και ο πρώτος ομιλητής και μετά θα ακούσουμε τον Δόκτωρα Ορτάκ. Ο κύριος Σάμπρη Μπαντάλ, ορίστε κύριε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ στο όνομα του Θεού και του Παγωνιού, κυρία Πρόεδρε και εσείς αγαπητοί φίλοι. Λέγομαι Μπεντεύ, θα ήθελα πρώτα να σας ευχαριστήσω όλους και να δηλώσω ότι είμαι ικανοποιημένο που βρίσκομαι εδώ και που μου δίνεται η ευκαιρία να ομιλήσω για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο λαός μου. Τεσσεράμιση χρόνια τώρα, όπου ο λαός μας ζει στους δρόμους, ε, χωρίς αιστείες. Δυστυχώς, λόγω ελλείψεως χρόνου, δεν θα μπορέσω να σας εξηγήσω ε, τα πάντα με ε, επαρκή λεπτομέρεια. Η τρομοκρατική βαρβαρική οργάνωση σκότωσε χιλιάδες ε, δικούς μας. Απήγαγε άλλες χιλιάδες και ανάγκασε σε εκτοπισμό άλλους. Αυτά τα πράγματα μα συνέβησαν. Πράγματα αδιανόητα. Αδιανόητα για τις σημερινές εποχές. Δεν σκέφτηκαν όμως την ανθρωπιά που θα έδειχνε η διεθνής κοινότητα. Διότι οι βάρβαροι αυτοί αντιμετώπιση των μελών της κοινότητας Γεσίδη αναχαιτίστηκε από την συνεργασία των δυνάμεων της Διεθνούς Συμμαχίας κατά του Ισλαμικού κράτους και κατάφεραν να εξαλείψουν το Ισλαμικό κράτος από το πρόσωπο της γης. Οι Γιασίδη δεν ήταν ποτέ πριν οπλισμένοι. Τώρα όμως χρειάστηκε να πάρουν τα όπλα και να ηγηθούν των δυνάμεών τους. Η γενοκτονία του 2014 και μετά από αυτήν εμείς οι Γεσίδη μέχρι τότε ήμασταν όλοι άμαχοι. Ποτέ δεν είχαμε εμπλακεί σε στρατιωτικές δραστηριότητες. Μετά όμως από το γεγονός εκείνο οπλιστήκαμε και εγώ ίδιος έγινα στρατιώτης στην υπηρεσία του λαού μου. Και μετά από αυτό χρειάστηκε να αναλάβω πολιτικές δραστηριότητες. Διότι σε αυτές πιστεύω και πιστεύω ότι η λύση του προβλήματος, των προβλημάτων που πλήττουν τον λαό μας, μπορούν ε, τα προβλήματα αυτά να λυθούν μέσω πολιτικών και ειρηνικών λύσεων. Και έχω κληθεί σήμερα για να μιλήσω για τις αξιώσεις του λαού μου. Αυτά που ζητεί ο λαός μου. έχουμε εκτοπιστεί και έχουμε γίνει πρόσφυγες στην ίδια μας την χώρα και ζούμε υπό απάνθρωπες συνθήκες. Λύση άλλη δεν βλέπουμε από την επιστροφή όλων των ανθρώπων μας στις αιστείες τους. Για να μπορέσει να γίνει αυτό σήμερα, φοβούμαι ότι εμείς είχαμε τα περισσότερα θύματα και παρόλα αυτά δεν αισθανόμαστε, και μάλλον γι' αυτό δεν αισθανόμαστε ασφαλείς στα χώματά μας. Σήμερα, εάν εκείνοι που βοήθησαν και συνεργάστηκαν με τον ISIS, με το Ισλαμικό κράτος, και έστρεψαν τα πυρά τους κατά τον Γεσίδη. Δεν μας αφήνουν τώρα να εγκατασταθούμε ξανά εκεί όπου είχαμε ζήσει. Όλες αυτές οι βάρβαρες επιθέσεις ωστόσο δεν είναι μόνο κατά του Σενγκάλ. Σήμερα ολόκληρη, ολόκληρη διοίκηση η κατάσταση επιδεινώνεται κάθε φορά που υπάρχει ένοπλη σύραξη, όπως για παράδειγμα στο Ιράκ. Στο Ιράκ υπάρχει, υπάρχει μία ένοπλη δύναμη που υπερασπίζεται τη χώρα. Στο Σενγκάλ όμως είναι 7. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω προβάλλοντας τρεις αξιώσεις των Γεσίδη του Σενγκάλ. Πρώτο, θέλουμε να επιστρέψουμε στις αιστείες μας, στη χώρα μας. Και οι χιλιάδες άνθρωποι που δεν εγκατέλειψαν ποτέ τα βουνά του Σιντζάς και οι πρόσφυγες και οι εκτοπισμένοι θέλουν και αυτοί να έρθουν στο Σενγκάλ και να μπορέσουν να ανοικοδομήσουν την περιοχή. Όπως συνεργαστήκαμε για να αντιταχθούμε στρατιωτικά στο Ισλαμικό κράτος, έτσι τώρα πρέπει να συνεργαστούμε για να χτίσουμε ξανά μια καινούργια ζωή, μαζί με την υποστήριξη βέβαια της περιφερειακής κυβέρνησης, ε, περιφερειακής κουρδικής κυβέρνησης του Ιράκ. Και πρώτα-πρώτα χρειαζόμαστε πολύ βασικά πράγματα. Σχολεία, ηλεκτρικό ρεύμα, χρειαζόμαστε υποδομή για ε, υδροδότηση. Δεύτερο, για να μπορέσουμε να χτίσουμε ξανά τη ζωή μας, ε, εμείς οι Γεσίδη, θα πρέπει να είναι εγγυημένη η ασφάλεια. Γιατί η ασφάλεια είναι αναγκαία για να μπορέσει κανείς να επιβιώσει. Την δε αυτοδιοίκηση του Σενγκάλ πρέπει να την αναλάβουν οι ίδιοι ΣΥΝΤΗ Και βέβαια θέλουμε ειρήνη μεταξύ ημών και των υπολείπων που ζουν στην περιοχή αυτή. Τρίτο, εγώ προέρχομαι από τη χώρα αυτή και θα ήθελα να πω ότι η ειρήνη αν γίνεται με το ζόρι δεν μπορεί να αποτελέσει βάση ε, για μακροπρόθεσμη ειρηνική συμβίωση. Γιατί η ειρήνη δεν μπορεί να προκύψει χωρίς δικαιοσύνη. Για να υπάρξει ε, βιώσιμη ειρήνη πρέπει να αναγνωριστούν οι γεσίδιοι και να αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ειρήνη. Αγαπητοί φίλοι, σας παρακαλώ και σας ζητώ να μας βοηθήσετε για να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας στην περιοχή μας. Και σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μας δώσατε σήμερα. Υπάρχει μια φυσική χρονική στέρηση γιατί περιμένουμε να τελειώσει η μετάφραση την οποία παρακολουθούμε. Δόκτωρο Τάκ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ, εξ ονόματος της οργανωσής μου στη Γερμανία, να σας ευχαριστήσω ένθερμα για αυτή τη πρόσκληση. Μετά από 4,5 χρόνια μιας γενοκτονίας ενός λαού στο Ιράκ και τη Συρία, χαίρομαι, παρόλο που με πονάει, που το θέμα αυτό εξεκολουθεί να είναι επίκαιρο και ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, εσείς δηλαδή. Αυτό μας χαροποιεί. Με χαροποιεί κυρίως το ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι εκτοπισμένοι, έχουν χάσει τους συγγενείς τους, τους συζύγους τους, τα παιδιά τους, μπορούμε να τους πούν, να, να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα ενδιαφέρονται για σας. Το 2014, όπως είπε και ο προλαλής σας, δεν θέλω να επαναλάβω τι έγινε, θέλω δύο-τρία πράγματα απλώς να αναφέρω. Εξ ονόματος λοιπόν της οργάνωσής μου από το 2014, πολλές φορές το χρόνο επισκεπτόμουν το Ιράκ. Και αυτό που ακούγαμε από τους Γεζίντι εκεί ήταν ειρήνη. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στη Γερμανία μπορούμε να αλλάξουμε τους, ε, τους νόμους, της, ε, την νομοθεσία, αλλά το μόνο που δεν μπορούμε να αλλάξουμε είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου την αξιοπρέπεια του ανθρώπου ή την αξιοπρέπεια ενός έθνους, ενός λαού. Από το 2014 προσπαθούμε με τον οργανισμό μου να έχουν αξιοπρέπεια και να ζουν με αξιοπρέπεια στη χώρα τους οι Γεζίντι. Σήμερα το πρωί είχαμε, κάναμε κάποιες διμερείς συζητήσεις και εκεί σε αυτές τις συζητήσεις έθεσα τα εξής θέματα ποια είναι τα σημαντικά για τους Γεζίντι. Όταν ήταν ε, το Ισλαμικό, το κράτος ακόμα εκεί, στην, ε, στη γη τους, είχαν ελπίδα ότι αυτή τη στιγμή νικηθεί το Ισλαμικό κράτος θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις αιστείες τους. Και δεν ήταν αδικαιολόγητη αυτή η ελπίδα, γιατί όταν έπεσε το Ισλαμικό κράτος, όλη η παγκόσμια κοινότητα και κυρίως οι Ευρωπαίοι αντέδρασαν όχι μόνο ανθρωπιστικά, ήταν καλό αυτό. Ήταν καλό που αντέδρασε η παγκόσμια κοινότητα. Και όταν ε, συζητώ εγώ με τους ανθρώπους αυτούς, μου λένε όταν νικηθεί το Ισλαμικό κράτος, εμείς θα επιστρέψουμε. Ε, θεωρητικά έχει νικηθεί το Ισλαμικό κράτος. Αλλά Όλοι επιστρέφουν στις χώρες τους, στη γη τους, μόνο οι γεζίντι δεν επιστρέφουν πίσω. Οι γεζίντι προσπαθούν πάντα να έχουν ε, διάλογο με την Ιρακινή κυβέρνηση και με την κουρδική κυβέρνηση. Εμένα η δική μου υποκειμενική άποψη είναι ότι αυτός ο διάλογος δεν είναι αμοιβαίος. Γι' αυτό δεν είναι καθήκον βέβαια μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του Κοινοβουλίου να το καταδείξει αυτό, γιατί οι μηχανισμοί που έχετε εσείς στα χέρια σας, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι διαφορετικοί σε σχέση με αυτούς που έχει η κοινωνία των πολιτών στα χέρια της. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρξει πολιτική πίεση προς και, και, τις, προς τις δύο κατευθύνσεις να, ρωτήσουμε, γιατί δεν μπορούν να επιστρέψουν οι Γεζίδοι στις αιστείες τους, στη χώρα τους. Γιατί ένα είναι ξεκάθαρο. Αν δεν έχουν μέλλον εκεί οι Γεζίδοι, θα πρέπει να γυρίσουν πίσω. Αν πλήττεται η αξιοπρέπειά τους, που γίνεται τώρα, συμβαίνει, θα πρέπει εδώ να τους υποδεχτείτε. Γιατί η γενικές ε, συλλογικές ε, διώξεις είναι άλλος ένας λόγος για να μην επιστρέψουν πίσω. Η αξιοπρέπεια λοιπόν του λαού μου δεν είναι απλώς, ε, δεν αποκαθίσταται όταν τους δώσετε μια μπουκιά ψωμί. Το θέμα είναι να μπορούν με περηφάνεια και με αξιοπρέπεια να ξαναχτίσουν τη χώρα τους. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό σημείο που όλοι εμείς από κοινού θα πρέπει να προωθήσουμε. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο. Ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει με περηφάνεια και με αξιοπρέπεια να επιστρέψουν στη χώρα τους. Εγώ έχω μιλήσει με πολλούς γεζίντι, γυναίκες και άντρες. Έχω μιλήσει με χριστιανικές ε, μειονότητες. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Αλλά όταν η πίεση είναι τόσο υψηλή, γιατί δεν λύνεται αυτή η διαμάχη, αυτή η σύγκρουση, τότε δεν μπορούν ήσυχα και χωρίς έννοιες να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ σε δύο εβδομάδες θα ξαναπάω πίσω. Και ελπίζω να μπορέσω να επισκεφθώ περιοχές που είναι, που ανήκουν στους Γεζίντι. Και επίση, πάλι μια υποκειμενική άποψη, ελπίζω ότι δεν είναι έτσι, αλλά οι περιφέρειες αυτές, τα σπίτια των, δράστων, των δραστών νομίζω ότι θα έχουν ε, ανοικοδομηθεί. Αλλά οι, οι υποδομές και οι περιοχές των θυμάτων σίγουρα δεν θα έχουν ανοικοδομηθεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλοι οι κρατικοί υπάλληλοι της κυβέρνησης υποχρεωτικά αναγκάζονται να επιστρέψουν στις περιφέρειές τους αν θέλουν να έχουν το μισθό τους. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό που υπάρχει αυτό το μέτρο. Αλλά στο Σενγκάλ, στις ε, περιφέρειες των Γεζίντι, αυτοί οι υπάλληλοι δεν υποχρεούνται να επιστρέψουν πίσω. Όπως είπε και ο προλαλή σα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχει ηλεκτρισμός, δεν υπάρχουν δρόμοι, σπίτια, έχουν όλα καταστραφεί. Η ειρηνευτική διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει. Και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ειρηνευτική διαδικασία μπορεί να επιτύχει μόνο αν το προσπαθήσουμε όλοι. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Okay, Σας ευχαριστώ. Έχουμε χρόνο, είναι σημαντικό το θέμα, έχουμε όμως λίγο χρόνο. Η ΕΔ είναι εδώ, έχουμε εκπρόσωπο. Δεν σας βλέπω καλά γιατί πολλά είπαμε εδώ για την πολιτική κατάσταση, για το θέμα της επιστροφής και των προβλημάτων που ακούσαμε. Ίσως θα ήθελα να ακούσω πρώτα την ΙΕΔ, προτού αναφερθούμε στην ανθρωπιστική κατάσταση. Ο κύριος Χάρισον, λοιπόν, εκ μέρους της ΙΕΔ, που είναι σαν την σαν το Υπουργείο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει η Πρόεδρος, για τους προσκεκλημένους. Ο κύριος Χάρισον έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας δίνετε το λόγο για να σας εξηγήσουμε τη δική μας ερμηνεία άποψη της κατάστασης στο Ιράκ και την περιοχή της Σίντζα. Ο συνάλφος θα μπορέσει να μπει σε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια για κάποια θέματα που μόλις έφυξαν οι αξιότιμοι προσκεκλημένοι σας. Καταρχάς, πολλά από αυτά που είπαν οι ομιλητές ε, α, αντιστοιχίζονται με την ε, δική μας, με τα δικά μας στοιχεία. Ε, το βασικό πρόβλημα στην περιοχή Σίντζα είναι η έλλειψη διακυβέρνησης, η έλλειψη διοικητική αρχή, η οποία πρέπει να προέρχεται από την κεντρική κυβέρνηση καθότι οι περιοχέ αυτέ. εν πάση περιπτώσει είναι υποδιαμάχη μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων και της ε, Ιρακινής αρχής λέει ο μιλητή. αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει διοικητική αρχή διακυβέρνησης για τα θέματα των πολιτών υπάρχουν τεράστια κενά στην, στην ασφάλεια. Υπάρχουν οι Ρακινές δυνάμεις, υπάρχουν ε, κάποιες ε, δυνάμεις ενόπλων μεταξύ των οποίων και Σιητών ε, που διαδραματίζουν ένα ρόλο εκεί και έχουν μια παρουσία και κάποιες ομάδες των κουρδικών δυνάμεων Εν μέρη βεβαίως όλα αυτά οφείλονται στο ότι δεν υπάρχει Υπουργείο Ιστορικών στο Ιράκ, η κυβέρνηση είναι ελλειπή. υπάρχει μια εσωτερική ενδοσκόπηση που τρέχει αυτή τη στιγμή στο Ιράκ. Το Σεπτέμβριο το Κοινοβούλιο του Κουρδιστάν, της περιφέρειας του Κουρδιστάν, συζητούν ακόμα για, για τον σχηματισμό κράτους, το οποίο είναι όμως μια διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί. Και η Τσιεζιντή, ο πνευματικό του ηγέτη από δεκαετία του 30, αν κάνω λάθος, πριν από λίγους μήνες εξέπνευσε και επομένω ε, βρισκόμαστε σε ένα κενό ηγεσία αυτή τη στιγμή μεταξύ διαφόρων ε, θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων. Στην καλύτερη περίπτωση το 10% του πληθυσμού έχει καταφέρει να επιστρέψει, αλλά άνω του 8% παραμένει σε στρατόπεδα και εντός της περιοχής του Κουρδιστάν για την πρόσβαση είχαμε εμπόδια τελευταία χρόνια και μέχρι πολύ πρόσφατα επί της αρχής επιτρέπεται η πρόσβαση αυτή τη στιγμή δεν οικοδομούνται εμπόδια βεβαίως υπάρχουν checkpoint σημεία ελέγχου από τους ενόπλους Σιήτες. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τεράστια κενά που υπάρχουν για την ασφάλεια της περιοχής μέσω του μέσου χρηματοδότησης για τη σταθεροποίηση του διεθνούς μέσου της διεθνούς κοινότητας συνεχίζουμε έργα στην περιοχή Σύντζα ε, ε, ε, ασκήθηκε πίεση από την, τα Ηνωμένα Έθνη στην ε, Διεθνή Συμμαχία, αλλά ακόμα και σε επίπεδο νοσοκομείων και σχολείων, ε, σημειώνουμε ότι ο πληθυσμός δεν επιστρέφει εκεί και αυτό μάλλον διότι υπάρχουν ακόμα ε, σημαντικά προβλήματα απειλής για την ασφάλεια. Επομένως, οι ντόπιοι ακόμα δεν αισθάνονται καθόλου ασφαλεί να επιστρέψουν. Δεν υπάρχει κάποια πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Ώστε να τους προσελκύσει πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια αλυσιδωτή βαθμία προσπάθεια για να έχουμε μια πιο επιχειρησιακά έτοιμη, αν θέλετε, προσπάθεια επιστροφής και επιπλέον επιβαρύνει το γεγονός ότι έχουμε συγκρούσει μεταξύ του ΠΚΚ και των ε, Ιρακινών δυνάμεων. Δύο κρούσματα είχαμε ε, στην βορειοανατολική Συρία πέρασαν τα σύνορα κάποιες δυνάμεις του ΠΚΚ και συγκρούστηκαν με τις Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και στην άλλη περίπτωση ήταν η YBS που είναι ομάδα των Γεζίντι που συγκρούστηκε με τις Συριακινές δυνάμεις. Μία, ένας από τους λόγους της μη επιστροφής είναι και το θέμα το ιδιοκτησιακό. Των τίτλων ιδιοκτησία. Ε, η ISIS κατέστρεψε τα περισσότερα από τα μητρώα που υπήρχαν και ε, επιστρέφουν τώρα όσοι επιστρέφουν ε, στα περιουσιακά στοιχεία που κατήχαν στο μεταξύ, στο μεσοδιάστημα, οι Σουνίτες γειτονέ τους και επομένως το ιδιοκτησιακό είναι θέμα σημαντικό. Η συμφιλίωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κανείς δεν έχει επιστρέψει μαζικά, δεν έχει ξεκινήσει από τη διαδικασία. Για ό,τι κάνει η Βρακή Ένωση υποστηρίζουμε το UNDP και το FSS, FFS μάλλον, με χρηματοδότηση και στην συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε κινητοποιήσει κάποιου χρηματοδοτικού πόρου τέλο πάντων για την περιοχή, λέει ο μιλητή με τεράστια ταχύτητα. Έχουμε και μια ερευνητική ομάδα των ΗΠΑ σχετικά με τα ε, εγκλήματα που διέπαρξε η Άσης ε, και έχουν ξεκινήσει στις έρευνες κάποιων μαζικών ε, τάφων στην περιοχή για αγνοωμένους που εξακολουθούν να είναι αγνοωμένοι επί των αγνοωμένων για κάποιους το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μάθουμε ποτέ την απάντηση, την αλήθεια αλλά έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια ε, για αυτήν την βασανιστική προσπάθεια να καταλάβουμε πόσοι ακριβώς ε, ε λείπουν, ε, πώς, πού κατέληξαν και πού βρίσκονται όσοι έχουν επιβιώσει. Ε, και φυσικά η έλλειψη υποδομή είναι αυτό που βλέπει κανείς άμεσα στην ε, περιοχή, αλλά μπορώ να σας πω ότι και στη Μοζούλη και αλλού στο Ιράκ ακριβώς τα ίδια βλέπουμε. Δηλαδή η όποια προσπάθεια συμφιλίωσης, ε, ειρήνευσης, σταθεροποίηση είναι εξαιρετικά πιο δύσκολη λόγω αυτού. Για να μην αναφερθώ σε ε, θέματα στεγαστικά. Αυτά είναι βέβαια της αρμοδιότητας της Ιρακινής Αρχής, λέει ο μιλτής, γνωρίζω ότι τα κράτη-μέλη αντιλαμβάνονται και ανησυχούν για τις καθυστερήσεις αυτής ε, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί στο Κουβέιτ πριν από ένα έντος. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε όμως την κατάσταση και μέσω των, των, των εργαλείων επικοινωνία που έχουμε στη διάθεσή μα ο πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. δώσω το λόγο, λέει η Πρόεδρο, στου υπολείπου, μία ερώτηση. Η ΕΚΟ είναι εκεί και όχι η Ωραία. Ε, ερώτηση λοιπόν. Μας λένε ότι η ISIS ε, είναι πλέον νητιμένη. Εξαφανίστηκε εν ολίγης. Κάποιοι από αυτούς κατέληξαν σε δυτικά χέρια, λέει η Πρόεδρος, και άλλοι στα χέρια της κυβέρνησης της Συρίας. Αλλά μία από τις ερωτήσεις της Νάντια Μουράτ δεν ήταν μόνο να καταλάβουμε πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αλλά να επιτύχουμε μια κάποια δικαιοσύνη για αυτούς που έχουν βιώσει και κατονόμασε έναν άνθρωπο που ήταν δημόσιος λειτουργός ως υπεύθυνο για, μαζική, για μαζικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και πριν από δύο εβδομάδες Συρία είχαμε άλλο ένα κρούσμα. Θα έχουμε κάποιες ε, πρωτοβουλίες για το Ιράκ, ε, για τέτοιου είδους κρούσματα. Η διεθνής κοινότητα θα οθήσει διεθνώς να υπάρξει μια συνέπεια να, συμμετάσχουν και οι Αμερικανοί και άλλοι. Αυτό θα συμβεί. Κοιτάξτε, η εντολή, η επίσημη εντολή συλλογής αποδείξεων και ενδείξεων ε, γιατί για τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να σας πω ότι για να ε, ξεκινήσει κανείς κάτι πρέπει να έχει αποδείξεις. Και έχουμε τα δύο εξή εκκρεμή. Πρώτον, από αυτούς που κατηγορούνται πόσοι είναι ακόμα ζωντανοί. Γιατί πολλοί από αυτούς έχουν σκοτωθεί στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ίσως αυτοί που έχουν επιβιώσει από τις επιθέσεις ή από την απελευθέρωση από τις Ιρακινές δυνάμεις, ίσως να έχουν διαφύγει προς Σύρια και να έμειναν στους τελευταίους θύλακες που είχε μέχρι πρόσφατα η ISIS εκεί στη Συρία. Πολλοί από αυτούς τους μαχητές τώρα ε, κρατούνται στην ε, βόρειο-ανατολική Συρία ή στο Ιράκ και πρέπει να καταλάβουμε ποιοι από αυτούς τους μαχητές κρατούνται ακόμα, είναι ζωντανοί, είναι υπεύθυνοι για αυτά τα εγκλήματα και μπορούν να διωχθούν. Τώρα για την συλλογή αποδεκτικών στοιχείων. Έχουμε πάρα πολλέ πληροφορίε που κυκλοφορούν, αλλά πρέπει να διασταυρωθούν και να επιβεβαιωθούν. Αυτό είναι προτεραιότητα για τα Ηνωμένα Έθνη και στο Ιράκ και ίσως και για τους ξένους μαχητές ή μάλλον τους μαχητές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ σκέπτομαι τα, την πρώη Λαβία, όπου γνωρίζαμε απολύτως καλά ποιοι ήταν οι δράστες αλλά δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε τα αποδεικτικά στοιχεία και αυτό χρειάστηκε τόσα πολλά χρόνια. Και επομένω ρεαλιστικά και στο Ιράκ έχουμε μια ακόμα πιο προβληματική κατάσταση. Ποιο έχει βιώσει, ποιο είναι ακόμα ζωντανό, αν θέλουμε δικαιοσύνη για αυτού που μπορούν ακόμα να διωχθούν και μετά να συλλέξουμε τα στοιχεία και να τα συνδέσουμε, να τα επιβεβαιώσουμε και να τα συνδέσουμε με του ανθρώπου αυτού. Και να βρούμε δικαστικού μηχανισμού στο Ιράκ ή μέσω ενό υβριδικού συστήματος που ακόμα δεν υπάρχει, μέσω του ψηφίσματος των ΗΕ 2379, ώστε να διωχθούν, να αποδοθούν δηλαδή ποινές στους υπευθύνους, στους δράστες. Τώρα αυτά που θα γίνουν στην πράξη είναι κάτι τελείως διαφορετικό και θα πρέπει να το δούμε στο άμεσο μέλλον. Πρόκειται για μια μακρά προσπάθεια δύσκολη, ακανθόδη, και η αποκατάσταση της αλήθειας, της ιστορικής αλήθειας θα πρέπει να λάβει μια μορφή ευρύτερη της διώξεως, της ποινική. Δηλαδή θα πρέπει τα γεγονότα να αποσαφινιστούν, που φαίνεται ίσως, ακούγεται ίσως λίγο δύσκολο, αλλά είναι απαραίτητο για μια συμφιλίωση. Θα πρέπει να έχουμε και μια προσπάθεια αποκατάστασης τη ιστορική αλήθεια του τι συνέβη σε εκεικμένες ζώνες και περιοχές ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διώξεω, ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποιου ανθρώπους μεταξύ των μαχητών ενδεχομένω που θα συνεργαστούν και που θα επιτρέψουν και στην κοινότητα των Γεζιντή να ξεπεράσουν το τραύμα τους. Η δίωξη είναι ένα τρόπο δικαιοσύνη, αλλά πρέπει να δούμε το θέμα ρεαλιστικά και η άλλη όψη της είναι να αποκαταστάσουμε τα τραύματα και κατά πόσο θα μπορέσουμε να διώξουμε πραγματικά τους υπευθύνους και τους δράστες γιατί ίσως να μην είναι πια εν ζωή. Um, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ να εξηγήσω στους προσκεκλημένους μας ότι είναι το τμήμα εκείνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι υπεύθυνο για την παροχή ανθρωπιστική βοήθεια. Θα μπορέσουν να απαντήσουν λοιπόν για θέματα άμεση βοήθεια. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσά κύριε για την παρέμβασή σα Λίγα λόγια για την ανθρωπιστική κατάσταση και τι έχουμε κάνει. Ως γνωρίζετε η ανθρωπιστική βοήθεια ήταν και μάλιστα από τις πρώτες και ήδη αρχίσαμε πριν από 4 ή 5 χρόνια στο Ιράκ με πάνω από 420 εκατομμύρια. που βέβαια στόχευαν στην ε, ανακούφιση των πιο ευάλωτων και μεταξύ αυτών βεβαίως των γεσίδη. Λίγα στοιχεία για το τι έχει γίνει και τι θα γίνει. Πρώτα, για τη γενετήσια βία. Οι γυναίκες των Γεσίδη βέβαια υπέστησαν τα πάνδυνα. Εμείς προσφέρουμε βοήθεια και προστασία για τέτοια θέματα τα τελευταία ε, δύο χρόνια στην περιοχή Σιντζάμπ όπου υπάρχει παρουσία Γεσίδη αλλά και όπου συγκεντρώνονται περισσότεροι από τους Γεσίδη που επιστρέφουν και για να μπω σε αυτά που είπε ο αξιότιμος προσκεκλημένος για τις θεμελιώδεις υπηρεσίες. Εκεί έχουμε καταβάλει τις μεγαλύτερες προσπάθειες για σύστημα στέγης και υγείας. Δυστυχώς ε, την προηγούμενη άνοιξη, λόγω των πλημμυρών αναγκαστήκαμε να ε, προσφέρουμε έξτρα ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών. Του τελευταίου μήνε και μετά από διάλογο με την κοινότητα των Γεσίδη και μετά από δικό του αίτημα, μετατρέψαμε την βοήθειά μας για μια βοήθεια διευκόλυνση αυτών που θα ε, διαβιώσουν εκεί τον χειμώνα και που αντιμετωπίζουν βέβαια τις βαριές συνέπειες ε, του βαριού χειμώνα σε υψηλό ε, επίπεδο, σε, δηλαδή σε επίπεδο, σε, σε μεγάλο ορεινό ύψος. Και ο ίδιο επίτροπο μα μας πήγε στο Ιράκ, επισκέφθηκε τη Σιντζά και ζήτησε βελτίωση της κατάστασης εκεί και μόλις προ λίγων ημερών, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επικεφαλή της ομάδος των δωρητών, δηλαδή όλοι οι δωρητέ που υποστηρίζουν τον Ερυθρό Σταυρό, κάθε χρόνο πηγαίνουμε κάπου ε, μαζί τους και εξετάζουμε την συγκεκριμένη περίπτωση και πήγαμε τώρα σε ολόκληρο το Ιράκ και ιδίω στο Βόρειο Ρακ, στην περιοχή των Κούρδων και των Γεσιντή, για να ζητήσουμε όλοι οι δωρητές να καταβάλουν έξτρα προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί να αντιμετωπιστούν τα κενά. Ένα μήνυμα έχω να μεταδώσω ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Στην στρατηγική μας λοιπόν για την ανθρωπιστική ανταπόκριση, HIP, Humanitarian κλπ. Η προσπάθειά μας δηλαδή για τις αρχές του 2019 και πρώτα για τις, μακρόχρο, για μακρόχρονες εκτοπίσεις, για τους μακρόχρονα εκτοπισμένους δηλαδή στο Βόρειο Ιράκ όπου βρίσκονται οι Γεσίδη και είναι η πρώτη μας προτεραιότητα αυτή και εκεί ε, δίνουμε ιδιαίτερα βοήθεια σε αυτούς που έχουν επιβιώσει της ε, βίας γενετήσιου χαρακτήρα. Και ένα άλλο θέμα, όπως ε, ε, έχουμε ξαναπεί, το ΕΚΟ δεν λειτουργεί μόνο του. Οι συνάδελφοί μου της ΔΕΦΚΟ, δηλαδή αυτοί που ασχολούνται με πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, εξετάζουμε τώρα με τους διαχειριστές των κονδυλίων πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ανοικοδόμηση του νοσοκομείου του Σιντζάλ και ζητούμε και από άλλες χώρες μέλη να συμβάλλουν. Δύο ακόμη σχόλια. Ευχαρίστως να συνεχίσουμε να συζητούμε ευθέως με την κοινότητα των Γεσίδη σε ό,τι αφορά την ανάλυση των αναγκών τους. Ευχαρίστως και μετά από την τωρινή συνάντηση να καθίσουμε μαζί, μας, μαζί σας και να δούμε, όπως γίνεται πάντοτε στην παρούσα Επιτροπή, ποιες άλλες ανάγκες έχετε. Και κυρία Πρόεδρε, ε, δεν είναι μονάχα για το Ιράκ, είναι και υπάρχει και η εμένη. Και θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την άμεση ανταπόκρισή του για την ανάγκη κινητοποίηση άμεση ανθρωπιστική βοήθεια για την Ιεμένη. Σα ευχαριστώ πολύ γιατί μπορέσαμε έτσι να ανταποκριθούμε με μεγάλη ταχύτητα. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή θα πάψει να συνεδριάζει το Κοινοβούλιο, να παραμείνετε σε επαφή με τη γραμματεία μας. Σας ευχαριστώ και εσάς για την εργασία που κάνετε. Θα επιστρέψω τώρα το μικρόφωνο. Ακούσατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μίλησε για την ανθρωπιστική βοήθεια και αν θέλετε διάλογο μαζί τους, να σκίσετε τώρα στις Βρυξέλλες, είναι καλή ευκαιρία. Αν κάποιος εξημών θα ήθελε να κάνει κάποιο τελικό σχόλιο, πριν να ολοκληρώσουμε το τμήμα αυτό της συνάντησής μας. Τώρα που ακούσατε τι κάνει η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μας ε, κοινοβουλευτική επιτροπή είναι κυρίως αρμόδια για ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή βοήθεια. Ακούμε όμως το μήνυμα που μας δίνεται ότι θέλετε να συζητήσετε, θέλετε να μιλήσετε και για την επιστροφή στις αιστείες σας. Κάτι που είναι πολύ φυσικό. Να φύγουν οι άνθρωποι δηλαδή από τους καταβλισμούς προσφύγων και αυτό μας απασχολεί και εμάς πολύ. Άρα θα μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό και στους συναδέλφους μας που ασχολούνται με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Άλλωστε περιλαμβάνεται και στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θέλετε να πείτε κάποια τελευταία λόγια, κάποιος εξ, εκ των δύο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα λόγια της και κυρίως για την υποστήριξη. Σας εύχομαι ε, κάθε επιτυχία στην περαιτέρω πορεία. Σας άκουσα ότι σήμερα είναι η τελευταία σας ε, συνεδρίαση. Είμαι πολύ ικανοποιημένο που αντιληφθήκατε το νόημα ε, του, μηνύματός μας. Είναι κυρίως πολιτικού χαρακτήρα. Όταν μιλείτε με στο Ιράκ, ζητήστε τους να έρθουν σε διάλογο μαζί μας και να μην μας παραβλέπουν και λαμβάνουν μέτρα χωρίς συζήτηση μαζί μας. Πρέπει να μιλήσουν με τους δικούς μας φορείς και τους δικούς μας ανθρώπους. Θα είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων αν μπορέσετε να το επιτύχετε αυτό. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκλησή σας και που μας επιτρέψατε να εμφανιστούμε ενώπιόν σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε εδώ, όπως σας είπα, υψηλούς αξιωματούχους και της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων και της ε, μονάδας ΕΚΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσαμε και εμείς το μήνυμα ως πολιτικοί και σας ευχαριστώ όλους και όλους που ε, ήσασταν σήμερα κοντά μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και να αντιληφθείτε παρακαλώ ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες σας. Θα επιτρέψω λίγα λεπτά για να μπορέσετε να αποχωρήσετε όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν και θα συνεχίσουμε. Θα δώσουμε ένα λεπτό στους ε, προσκεκλημένους μας για να μπορέσουν να αποχωρήσουν. Okay, colleagues, can I ask those who are leaving to leave because... Παρακαλώ όσοι επιθυμείτε να αποχωρήσετε, να αποχωρήσετε γιατί θέλουμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Και δεν θα... Α, βλέπω ότι ο Γκέρχολτ είναι παρόν. Τι ωραία, πολύ καλά. Ε, συμπίπτει απολύτως χρονικά. Παρακαλώ λοιπόν, εφόσον αποχωρούν οι ε, προσκεκλημένοι μας, ε, να προχωρήσουμε στο υπαριθμό 9 Πρόκειται για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών στη Σενεγάλη για τις προεδρικές εκλογές της 24ης Δευτέρου. Είχα και εγώ την ευκαιρία να πάω και ήταν και η πρώτη μου αποστολή παρατήρησης εκλογών. Τόσο το καλύτερο, διότι είχαμε μια θαυμάσια επικεφαλή στην κυρία Βαλενσιάνο, ε, πραγματική, εξαιρετική και με ε, πολύ ηγετικό ταλέντο. Και Μιλήσαμε και πριν για την Άντια Μούρατ και θυμούμε πόσο εργάστηκες για την Άντια Μούρατ και την βράβευσή της. Η Έλενα Βαλενσιάνο λοιπόν ήταν η επικεφαλής της αποστολής μας. Κοντά μας είναι και ο Στέφαν Γκέρολντ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Σενεγάλη τις ημέρες που ήμασταν εκεί. Ε, θα είναι σύντομη η ανταλλαγή απόψεων για τα πρακτικά περισσότερο. Κυρία Βαλενσιάνο, λοιπόν. Ευχαριστώ. Πραγματικά ήταν ικανοποίηση να συμμετάσχω στην ε, αποστολή αυτή παρατήρηση εκλογών στη Σενεγάλη. Σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαντική χώρα για ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο. Η εκλογική διαδικασία ήταν ήρεμη, διαφανής με σημαντική κινητοποίηση του εκλογικού σώματος, παρότι καταφέραμε να διακρίνουμε μία ατμόσφαιρα σημαντικής έλλειψης εμπιστοσύνης, χάσματος μεταξύ της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της α, αντιπολίτευσης, της πολυσχηδούς αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση επανεξελέγει με άνω του 58% και αυτό κατέληξε σε διάφορες νομοθετικές ε, προσαρμογές, τροποποιήσεις, το οποίο ο πληθυσμός δεν το υπεδέχθη καθόλου θερμά. Και προσπαθώντας να αναπτύξει ο κυβερνητικός ε, σχηματισμός ε, μια πολιτική συνένεση. Υπέβαλε και προτάσεις, οι οποίες απέρριψε η αντιπολίτευση, η προεκλογική εκστρατεία καθεαυτή. Ήταν αρκετά ελεύθερη και ήρεμη, με απόλυτη ανισορροπία βέβαια μεταξύ οικονομικής δυνατότητας και ισχύω ε, κυβερνητικής και αντιπολίτευσης. Αλλά, η πάση περιπτώσει, οι πολιτικές δυνάμεις διεξήγαγαν τις ε, προεκλογικές συναντήσεις ε, και την εκστρατεία τους εν ειρήνη και ηρεμία. Η ατμόσφαιρα λίγο άλλαξε όταν, άλλαξε όταν ο πρώην πρόεδρος Γκουάντε άσκησε πίεση για να μποϊκοτάρει τις εκλογές το οποίο δεν κατόρθωσε η, κοινωνία της Ενεγάλης δεν ήταν, δεν ήταν καθόλου διατεθειμένη για αντιπαράθεση και έτσι ο Γκουάντε ούτε κατόρθωσε τίποτα ούτε υποστήριξε άλλον υποψήφιο. Ο πρόεδρος Μακισάλ έλαβε το σχεδόν 59% με σχεδόν το σύνολο του εδάφους ε, κέρδισε τις εκλογές με μια εκλογική πλατφόρμα με πάρα πολλά κόμματα από το φιλελεύθερο μέχρι το σοσιαλιστικό κόμμα. Δηλαδή μια εκλογική πλατφόρμα ευρύτατη, ευρύτατου του φασμάτος. Και αυτό το επράγησαν οι εκλογείς, το εκλογικό σώμα. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητος ο διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, διότι υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας που δεν πρέπει να υπάρχει σε μια δημοκρατία που είναι εγκαθιδρυμένη όπως αυτή της Σενεγάλης. Είναι η ενδέκατη φορά που ε, ψηφίζουν οι Συνεγαλέζοι. Είναι μια χώρα πρότυπο, παράδειγμα για το υπόλοιπο της ε, περιοχής και της Υπήρου. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσει λοιπόν στην κατεύθυνση αυτή. Μας υπεδέχτησαν πολύ θερμά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, νομίζω ότι υπάρχει και μια δουλειά πολύ ενδιαφέρουσα που πρέπει να γίνει από σε αφρικανικών ενώσεων που ήταν παρούσες εκεί και με τις οποίες ε, συμμεριζόμαστε το σύνολο στην πραγματικότητα των συμπερασμάτων παρατηρήσεων μας. Επομένως, εκλογική διαδικασία καλή, προοπτική συνέχισης συνεργασίας της ενεγάλη και αναγκαιότητα, ξαναλέω, επανεκκίνηση διαλόγου με την αντιπολίτευση και την ε, επανεκλεγήσα κυβέρνηση. Ευχαριστώ, Λίντα. Θα μιλήσω γερμανικά. Να πω ότι ήταν ιδιαίτερες αυτές οι εκλογές. Ε, εγώ έζησα κάποια χρόνια στη Σενεγάλη και γι' αυτό η αποστολή αυτή ήταν πραγματικά ιδιαίτερη, είχε ιδιαίτερη σημασία. Η κοινοβουλευτική μας αντιπροσωπεία αποτελεί το από πέντε συναδέλφους του Κοινοβουλίου συν την ε, Έλενα Βαλενσιάνο, την, ε, το αφεντικό μας που έκανε πραγματικά εξαιρετική δουλειά και πάλι την ευχαριστώ θερμά γιατί ήταν πραγματικά συναρπαστική η ηγεσία που έδειξε. Ε, να ευχαριστήσω επίσης το σύνολο της ομάδας έκανα πραγματικά πάρα πολύ καλή προετοιμασία και η διαμονή μας στη Σενεγάλη ήταν πραγματικά απρόσκοπτη και γι' αυτό νομίζω ότι οδηγηθήκαμε τελικώς και σε επιτυχία στην αποστολή αυτή. Όπως είπε και η Έλενα Βαλενσιάνο, δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα. Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη επιτυχώς υπό καλέ συνθήκε. Νομίζω ότι ο λαός της Σενεγάλης είναι ο πρώτος που κέρδισε από, αυτές τις, από αυτή την διαδικασία. Μία μικρή προσθήκη να κάνω στο προσκήνιο, ευτυχώς. Δεν, υπήρξε, δεν υπήρξαν προβλήματα στην ε, εκλογική διαδικασία ε, παραχάραξης ή συγκρούσεων. Ε, υπήρξαν βεβαίως, υπήρξε ένα μικρό κρούσμα με δύο ε, θανάτους, δύο θύματα. Ε, ξέρουμε ότι οι αστυνομικές αρχές και η εισαγγελία ερευνούν την, το, την περίπτωση αυτή, αλλά δεν υπήρξαν σειράξεις, ήταν ειρηνικές αυτές οι εκλογές και μπορούσαμε να κάνουμε και κριτικά σχόλια χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν επιθετικές συμπεριφορές. Τώρα, ένα έτσι κάπως αρνητικό, γκρίζο σχόλιο. έπρεπε να αναγνωρίσουμε ότι η ε, εκλογική επιτροπή δεν είχε ε, προετοιμαστεί επαρκώς. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σύνηθες, αλλά επειδή ήμασταν και στην καταμέτρηση παρόντες, μας φάνηκε ότι χωρίς να υπάρχει κακοπιστία, αλλά επειδή υπήρχαν ε, ελλείψεις σε γνώση και σε προετοιμασία, η ε, Φορευτική Επιτροπή δεν έκανε πολύ καλή δουλειά. Αυτό το παρατήρησαν και άλλες αποστολές παρατηρήσεις εκλογών που ήταν παρούσες. Η εκπαίδευση η κατάρτιση αυτών που πρέπει να οργανώσουν την εκλογική εκστρατεία είναι απαραίτητη, είναι εκ των για να μπορεί έτσι και εθνικά αλλά και σε διεθνέ επίπεδο να αναγνωριστούν να αναγνωριστεί ότι οι εκλογές έγιναν σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές. Επίσης, άλλο ένα προβληματικό σημείο ήταν η... Ε, το σημειώσαμε και ε, παρά τις ε, διαφορετικές απόψεις του, ε, του πρέσβη μας, είδαμε έναν μεγάλο κατακαιρματισμό. Το πολιτικό σύστημα έχει δύο βασικά πολιτικά κόμματα στη Σενεγάλη. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα υποστήριξε στο τέλος των εκλογών τη συμμαχία που θα δημιουργούσε ο νέος πρόεδρος, αλλά δεν είχε δικό του ε, υποψήφιο, τουλάχιστον ε, την ημέρα των ε, εκλογών. Ε, αυτές οι εξελίξεις βέβαια είναι παρόμοιες και σε άλλες χώρες, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι μια σωστή δομή των, του πολιτικού συστήματος θα γίνει μέσω κατευθυντηρίων γραμμών. Θα ήταν καλό να γίνει μια σχετική ε, συζήτηση. Ο πρόεδρος ε, Μαρκισάλ ε, επανεξελέγει. Δεν υπήρχαν αμφιβολίες για την νίκη του. Έχει σημαντικά καθήκοντα να αναλάβει. Και βεβαίως και ο πολιτικός κόσμος της Σενεγάλης έχει σημαντικά καθήκοντα να αναλάβει για την ανικοδόμηση του πολιτικού συστήματος. Αυτά από μένα, πρόεδρε, και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και τους δύο. Είναι κάποιος ακόμη εδώ από την ΕΙΕΔ, ο Ρικάρντο Τσελέβη, θα μας ενημερώσει από τις εξελίξεις από την ολοκλήρωση της αποστολής και μετά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ένα ένθερμο ευχαριστώ στην Έλενα και στο Στέφαν, αλλά και σε εσά για την υποστήριξη στην παρατήρηση των εκλογών. Ήταν πραγματικά παραδειγματική αποστολή, συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν στο ύψιστο επίπεδο. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και μπρος. Η αποστολή από κοινού και με την Έλενα προσπαθεί να ορίσει μια επίσκεψη μάλλον τον Ιούνιο. Η, επίσης δουλεύουμε πάνω στην τελική έκθεση που θα περιλαμβάνει και κάποιε συστάσει. Οπότε τον Ιούνιο η Έλενα θα επιστρέψει με ένα τμήμα της ομάδας για να συζητήσει τις ε, ε, συστάσεις μας με τις συναγαλλικές αρχές. Και θα γίνουν επίσης και κάποιες στρογγυλές τράπεζες συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να ξεκινήσει η δουλειά για την εφαρμογή των συστάσεων. Αυτό γίνεται συνήθως βέβαια. Ελπίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εμπλακεί και στην μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των συστάσεων, γιατί συμβάλλουν στην βελτίωση του ε, εκλογικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί η Σενεγάλη. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Έλενα. Just for the record. Um, ναι, Πρόεδρε. Ήθελα να υπογραμμίσω την ε, σημασία που έχει η δουλειά αυτή των αποστολών παρακολούθησης εκλογών δηλαδή και τις σημασίες που έχει η συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου, της ΙΕΔ και της Κομισιόν. Το προσωπικό της ΙΕΔ και της Επιτροπής έχει ένα υψηλότατο επίπεδο προετοιμασίας, εξειδίκευσης, ικανότητας και δυνατότητας ανάλυσης σε μια τρίτη χώρα, τρίτη χώρα, με συγχωρείτε, πρόκειται για ανθρώπους που πραγματικά αξίζει τον κόπο να τους γνωρίσει κανείς τους ίδιους και τη δουλειά τους και θεωρώ θεμελίωδη σημασία στη δουλειά αυτή. Όπως λέει ο Στέφαν, η συνεργασία αυτή ήταν εξαιρετική και όπως λέει και ο Ρικάρντο, πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε, όταν συνεργαζόμαστε, συνομιλούμε με τους Σενεγαλέζους για τη βελτίωση του πολιτικού του συστήματος, πέραν των εμπειρογνωμόνων και των ειδικών των τεχνικών, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν, να είναι παρόντες οι βουλευτές. Τώρα, ε, ε, κάποιοι δεν είναι πλέον μέλη. Αυτοί που είναι και συμμετέχουν και συνεχίζουν, πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις αποστολές, να είναι παρόντες, γιατί είναι σημαντικό να δίδεται επιφάνεια σε αυτή την προσπάθεια, να είναι πιο εμφανής. Ευχαριστώ λοιπόν Στέφαν, ευχαριστώ Λίντα. Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ σένα Ελένα και επαναλαμβάνω αυτό που είπες για τη σημασία ε, να συμμετέχουν και πολιτικοί, διότι η Σενεγάλη είναι διαφορετική από την Ισπανία, την Γερμανία, αλλά έχει και ομοιότητες. Έχουν παρόμοιες οργανώσεις, έχουν δασκάλους που ε, λειτουργούν τα σχολεία στα οποία γίνονται, γίνεται οι ε, εκλογές και επίσης ανθρώπους που ε, καταμετρώνουν ψήφους κλπ. Βλέπω και την Μπιζίτ Μπατάγ, ε, βλέπω και ε, τους άλλους ανθρώπους, ε, θαυμάσιους ανθρώπους της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων που εργάζονται σκληρά και έχουμε και πολλούς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εργάζονται για τα θέματα αυτά με πολύ συστηματικό τρόπο και ελπίζω και ε, στο επόμενο κοινοβούλιο να συνεχιστεί αυτό. Προσκαλέσαμε τους ανθρώπους του ΔΕΚ στις 6.30. Αν ε, τα γνωρίζετε αυτό όμως, αν είστε εύκαιροι θα έρθετε. Και βεβαίω αυτό ισχύει και για τους συναδέλφους της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων. Ε, τώρα έχουμε να μιλήσουμε για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών στην Ιγυρία. Κένια, υπά, ήταν λάθο. Ε, είναι το θέμα λοιπόν, λοιπόν υπάρχουν 10. Αποστολή εκλογική παρατήρηση στην Ιγυρία στις 23 Φεβρουαρίου 2019. Αυτή η αποστολή ήταν δύσκολη, δεν θα πω τίποτε περισσότερο, γιατί η Μαρία Αρενά ε, ήταν ε, μέλος της ε, αντιπροσωπής αυτής. Δύσκολη λοιπόν ε, αποστολή παρατήρηση εκλογών, οι οποίε εκλογέ αναβλήθηκαν λίγε ώρε πριν να ανοίξουν οι κάλπε. Χαίρομαι που έχουμε κοντά μα τη Μαρία Αρενά, που ήταν η επικεφαλή, και τον Σαντιάγο Φίσα, που ήταν ε, επικεφαλή τη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Μαρία Αρενά, γνωρίζω ότι ήταν δύσκολη ε, η αποστολή σας αυτή και αν μπορείτε να μας πείτε τι συνέβη και τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε. Ευχαριστώ πράγματι. Δύσκολες και περίπλοκες εκλογές. Και μιλούμε για 84 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Ε, ήδη είναι δύσκολο αυτό να οργανωθεί και σε μια χώρα επίσης δύσκολη. Με ε, διέρεση βορρά-νότου, με υποψηφίους που καμιά φορά ήταν δύο μουσουλμάνοι υποψήφοι ενώ κανονικά εναλλάσσονται ε, ανάμεσα στον ε, μουσουλμανικό βορρά και στον χριστιανικό νότο ε, ή δύσκολο το πλαίσιο των εκλογών αυτών και μάλιστα τόσο περίπλοκο που την ίδια την ημέρα της εκλογής αποφάσισαν να αναβάλουν και τις προεδρικές εκλογές, την προεδρική εκλογή δηλαδή, ταυτόχρονα όμως και τις τοπικές, δηλαδή για τους κυβερνήτες επαχιών ή διοικητικών διαμερισμάτων. Και ε, μετά από την προεδρική εκλογή που επιβεβαίωσε τον πρόεδρο βουάρι του κόμματος ΑΠΣΕ που κέρδισε τις εκλογές και μάλιστα με ευρεία διαφορά. Και οι ενδεχόμενες αμφισβητήσεις δεν θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τελικώς το αποτέλεσμα των εκλογών το αποτέλεσμα το οποίο έγινε αποδεκτό και από τον κόσμο, από το κοινό δηλαδή. Πιο περιπλοκή ήταν η κατάσταση για την εκλογή των κυβερνητών με την έννοια όπου κάθε πολιτεία έχει εκπροσώπηση άπεσε και 5 που είναι πολύ εγγύς και μπήκαν σε μια λογική αμφισβητήσεων ενστάσεων για την εκλογή των κυβερνητών Υπήρχαν και οργανωτικές δυσκολίες με αναβολές για έξι διαφορετικές πολιτείες που χρειάστηκε να οργανώσουν εκλογές για αργότερα. Με επεισόδια βίας σε ορισμένες πολιτείες, αλλά και με επεισόδια όπου όλη η συνέχεια των αποτελεσμάτων των εκλογών και ιδίω για τα κέντρα καταμέτρησης, εκεί η διαδικασία δεν ήταν διόλου διαφανής και υπάρχουν επομένω πολλές προσφυγές που έχουν κατατεθεί ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένη εκλογής. Πρόκειται για μια χώρα ε, εύθραυστη σε ό,τι αφορά την δημοκρατική δομή της. Έφραστη διότι υπάρχουν και σημαντικά διακυβεύματα ασφαλείας σε ολόκληρη την χώρα και κυρίως στο βόρειο-ανατολικό τμήμα όπου δράει η οργάνωση Μπόκο Χαράμ, είναι η περιοχή του Σαχέλ. Έφραστη επίσης διότι υπάρχουν και άλλα διακυβεύματα όπως ε, η θέρμανση του κλίματος αλλά και σημαντικές διαμάχες ανάμεσα σε αγρότες και κτηνοτρόφους στο κέντρο της χώρας. Συγκρούσεις οι οποίες παίρνουν και εθνοτικό χαρακτήρα διότι οι κτηνοτρόφοι είναι περισσότερο μια εθνότητα μουσουλμανική ενώ οι ε, ε, γεωργοί είναι οι καλλιεργητές δηλαδή περισσότερο από χριστιανικές εθνότητες του Νότου και είναι μια ε, σύγκρουση και οικονομική που τελικώς ενδύεται τον μανδύα της εθνοτικής σύγκρουσης και θρησκευτική. Και ένας τρίτος παράγων που συνδέεται με το πετρέλαιο και όλη την σχετική διαφθορά γύρω από την εκμετάλλευση των πόρων αυτών. πάλι του νότιου μέρους όπου βρίσκονται οι εκμεταλλεύσεις του πετρελαίου και όπου οργανώνεται σημαντική κλιματική δραστηριότητα. Συντάσσουμε μια τελική έκθεση την οποία θα καταθέσουμε τον Ιούνιο στην επίσκεψη που θα κάνουμε πάλι εκεί και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πολύ ακριβείς συστάσεις για τις επόμενες εκλογές του 2021 διότι αυτό το εύθραυστον 2023 νομίζω, 2023, με συγχωρείτε, 2023. Αυτός ο έφραστος χαρακτήρας θα ενισχυθεί ενδεχομένως μέχρι το 2023 και θα πρέπει οι συστάσεις αυτές να ληφθούν υπόψη από την νέα κυβέρνηση. Συνεργαστήκαμε καλά και με την Επίρρηση Εξωτερικών Δράσεων και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την αντιπροσωπεία που έκαναν αξιοθαύμαστη εργασία οργανώνοντας συναντήσεις με τους διαφόρους φορείς και της κοινωνίας των πολιτών και του ΑΙΝΕΚ e και των άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται επί τόπου και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και με συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία Επιτόπου, ώστε να μπορέσουμε με την εκθεσή μα να προχωρήσουμε δυνατόν συντομότερο. Για παράδειγμα, και με τι συστάσει που διατυπώθηκαν αμέσω μετά τι εκλογέ, ώστε να γίνουν η βάση για ένα ε, εθνικό διάλογο να αρχίσει ένας προβληματισμός λοιπόν για τις επόμενες εκλογές όσον αφορά τις ελλείψεις που διαπιστώσαμε στο εκλογικό σύστημα της Νιγηρίας. Η συμμετοχή υστερούσε απέναντι και στην προηγούμενη και υπάρχει και ε, μειωμένη εκπροσώπηση γυναικών, εκπροσώπηση ακόμη πιο χαμηλή από άλλες φορές είναι λοιπόν δύο θέματα τα οποία είναι σημαντικό να τεθούν όταν μιλούμε για σύστημα, δημοκρατικό σύστημα το οποίο να μην αποκλείει κανένα. Άρα, ε, ε, ελλείψη δημοκρατικότητα του συστήματο και έλλειψη εκπροσώπηση ή απαρκού εκπροσώπηση των γυναικών. Ορίστε, αυτά ήταν ε, όσα ήθελα να σα πω. Ευχαριστώ. Εσεί, κύριε Φίσα. Θα μιλήσω στα Ισπανικά. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Μαριά εξαιρετικά περιέγραψε το κλίμα και την κατάσταση. Νομίζω ότι επίσης ε, κάναμε μια εξαιρετική δουλειά. Ήταν δύσκολες εκλογές, περίπλοκες. Εγώ ήμουν ο προηγούμενος επικεφαλής παρατηρητής στις προηγούμενες δηλαδή εκλογές και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες της χώρας αυτής που είναι πολύ μεγάλη και με τάσεις αύξησης του πληθυσμού ε, τεράστιες με διάφορες εθνικές ομάδες ε, και πολύ σημαντική ποσόστοση μουσουλμάνων, ε, περίπλοκη λοιπόν χώρα, με οικονομία βασίζεται στο πετρέλαιο και οικονομία σημαντική. Δεν θα επεκταθώ σε αυτά, αλλά απλώς θα πω ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε κάπως... Ε, δεν μπορούμε να, να ε, παρασταθούμε στην, στην ημέρα των εκλογών. Δηλαδή, εμείς στην περίπτωση τη δική μας τότε, ε, μας έδιωξαν στις 2.30 το πρωί της ημέρας ε, των ξημερωμάτων της ε, ημερομηνίας των εκλογών. Μετά ανεβλήθη η εκλογή, δεν βρίσκαμε τους συναδέλφους για να ξαναπάμε κτλ. Ε, ε, εξεπλάγιν εγώ κάπως ε, από τη στάση που κράτησε η ΑΙΝΕΚ που είχε τέσσερις, τέσσερα χρόνια να διοργανώσει τις εκλογές και στο τέσσερα το απόγευμα της προηγουμένης μας ε, υποδέχθηκαν στην ΙΝΕΚ, ε, τους ρωτήσαμε, όλα πάνε καλά, μας έλεγαν, αύριο θα έχουμε εκλογές, όλα καλά, στις 4 το απόγευμα της προηγουμένης. Και μετά τα ξημερώματα ανέβαλαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι ε, τεχνικός μιλώντας δεν ήταν όλα έτοιμα, σε καμία περίπτωση. και κάποιοι σκέφτηκαν ότι πίσω από αυτό κρυβόντουσαν κάποιες έτσι άλλες πολιτικές ή στρατηγικές τοποθετήσεις αναβολής των εκλογών αυτών. Εν πάση περιπτώσει αναφερθήκατε, αναφέρθηκαν συνάδελφοι σε μεγάλη εποχή στην Ιγερία απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Πρέπει κανείς να πάει με τα πόδια. Σκεφτείτε λοιπόν αν είναι για μα ενοχλητικό. Φανταστείτε τους Νιγηριανού πρέπει να περπατήσουν χιλιόμετρα για να πάνε να ψηφίσουν και στην περίπτωση της δικής μας παρατήρησης περπάτησαν τα χιλιόμετρα και μετά τους είπαν δεν μπορείτε να ψηφίσετε. Δηλαδή, εάν είναι να κάνει κάνει τέτοια προσπάθεια ε, με πενιχρά μέσα για να πάει να ψηφίσει και του λένε δεν μπορεί, την επόμενη δεν πάει. Είναι προφανέ λοιπόν ότι είναι δύσκολε συνθήκε μία από τις ε, ε, συστάσεις που εμείς είχαμε υποβάλει την προηγούμενη φορά ήταν μάλλον προηγουμένως έπρεπε να εγγραφούν το πρωί, το ίδιο πρωί οι πολίτες στο σπίτι τους, λέει ο για να μπορέσουν να ψηφίσουν το απόγευμα. Δηλαδή, αν ήταν στην Ευρώπη να κάνουμε αυτό το πρωί χωρίς οχήματα, με τα πόδια, να πάμε να εγγραφούμε για να γυρίσουμε σπίτι και να πάμε μετά να ψηφίσουμε το απόγευμα, αναρωτιέται κανεί τι θα συνέβαινε. Δηλαδή, πρέπει κανείς και να αναγνωρίσει τον ενθουσιασμό των ε, πολιτών της Νιγηρίας για την δημοκρατία με όλα αυτά που υφίστανται για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Πάντω. υπήρχε δυνατότητα εγγραφή και ψήφου με αυτά που σας είπα. Εν τόσοι οι τεχνικές δικαιολογίες που χρησιμοποιήθηκαν θα δούμε αν είναι αληθής ή όχι. Αλλά δεν μιλάμε για μια φτωχή χώρα. Δεν μιλούμε για μια φτωχή χαμένη χώρα. Μιλούμε για μια από τις ισχυρότερες, πλουσιότερες χώρες της Αφρικής, της Αφρικανικής Επίρου. Είναι δυνατόν να μην έχει τα μέσα στη διαθεσή της για να διοργανώσει μια εκλογική διαδικασία που το απόγευμα της προηγουμένης μας διαβεβαίωναν ότι καλός έχει και ότι θα διεξαχθεί μια χαρά. Και όταν εγώ ήμουν επικεφαλής αποστολής, ε, τουλάχιστον αυτό το έκαναν, είχαν την, την λεπτότητα, αν θέλετε, να το κάνουν εντός μια εβδομάδα, μιας εβδομάδας την αναβολή. Ε, σε αυτή την περίπτωση την έκαναν την, την αυτή ημέρα, την ίδια μέρα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις και κενά. Αλλά θα ήθελα να συγχαρώ τη Μαρία γιατί πραγματικά μιλούμε για μια δύσκολη, δύσκολη κατάσταση, περίπλοκη, ε, που μεταξύ περιφερειαρχών εκεί κυβερνητών ε, επαρχείων ήταν και λίγο εκρηκτική σε κάποια επίπεδα, όμως ε, νομίζω ότι έγινε εξαιρετική δουλειά συνολικά. Uh, Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και για αυτό το θέμα που θίξατε για την τεχνολογία. Ε, εμένα πάντα με ενοχλεί λίγο η υπερβολική χρήση τεχνολογίας στις ε, εκλογές. Σε πολλές χώρες ε, δεν λείπει η υπερβολική τεχνολογία, λείπουν μολύβια για να μετρήσει κανείς τις ε, ψήφους. Οπότε ας απλουστεύσουμε λιγάκι τα πράγματα. Ε, βέβαια δεν ξέρω, η, η θα μπορούσε κάτι να μας πει από αυτού. Δεν ξέρω αν οι άλλοι συνάδελφοι θέλουν κάτι να πούν. Ο Τζόρτζο Χόκκιν. Όχι. Α, θέλεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για τις αναφορές, όντως αυτά που είπατε, αυτά συνέβησαν. Εγώ πήγα στο Λάγκος και εκεί ως έκπληξη αναβλήθηκαν οι ε, εκλογές αλλά δεν το καταλάβανε όλοι. Ε, και στην ε, τοπική εκλογική επιτροπή οι γραμματέας ήταν εκεί και όλα τα μέλη που έπρεπε να είναι εκεί και ήταν εκεί, ήταν Ε, μας είπανε, ρωτήσαμε πού είναι όλα τα, όλο το υλικό των εκλογών, μας στείλανε στην κεντρική τράπεζα που είχε μόνο κανένα αστυνόμους. Μας είπανε δεν μπορούμε να σα αφήσουμε, δεν είναι κανένας μέσα. Μετά πήγαμε στις τοπικές αρχές, σε έναν από τους δημάρχους και μας είπε ναι το, το βράδυ ε, θα έρθουν 550 ε, υπάλληλοι για να βοηθήσουν, μάλλον και αυτοί θα εξεπλάγησαν ιδιαίτερα. Μείναμε, μείναμε εκεί λοιπόν, ε, μοιραστήκαμε στους ε, στα διάφορα εκλογικά κέντρα. Ήταν λίγο περίεργο αυτό το σύστημα και ε, λιγάκι μας, ε, μας άγχωσε, μας εκνεύρισε. Και τα μικρότερα κόμματα, τους εκλογικούς τους αντιπροσώπους, τους είχαν πληρώσει, ενώ τα δύο μεγάλα κόμματα όχι. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Τα μικρά κόμματα Μα είπαν αν γίνουν οι εκλογέ σε μια εβδομάδα, ε, οι δικοί μα ε, θα είναι ε, στο σπίτι του και δεν θα μπορούμε πάλι να του ξαναδώσουμε λεφτά αν δεν έρθουν για να, γίνει τώρα, να γίνουν τώρα οι εκλογέ. Ενώ για τα μεγάλα κόμματα δεν ήταν πρόβλημα αυτό. Στι 4 η ώρα κάναμε τη συζήτηση με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Μα είπαν όλα καλά, όλα έτοιμα και λίγες ώρες μετά ακούσαμε ότι αναβάλλονται οι εκλογές. Προφανώς αυτά που δεν ε, ήταν έτοιμα ε, μετά από τέσσερα χρόνια δεν θα ετοιμάζονταν μέσα σε λίγες ώρες. Ήταν κρίμα. Γιατί χρειάζεται δημοκρατικές σχέσεις αυτές, αυτή η χώρα για να λύσει τα προβλήματα που έχει και είναι πολλά. Τα είπε πολύ καλά η κυρία Ρένα. Είναι μια χαμένη ευκαιρία. Τώρα αν δούμε ε, εκ των υστέρων τις εκθέσεις, νομίζω ότι θα φανεί και εκεί όλη αυτή η αταξία στις, ε, για τις κυβερνητικές τοπικές εκλογές που ίσως είναι πολύ πιο σημαντικές γιατί αυτοί οι τοπικοί άρχοντες είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη στα χέρια τους τελικώς. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει πραγματική τακτική διαδικασία για τις εκλογές, οπότε και εγώ περιμένω εναγωνίως να δω τι θα προκύψει. Η Μαρία Ρένα φαντάζομαι ότι θα μας ενημερώνει σχετικώς φαντάζομαι ότι θα γίνουν εκλογές κάποια στιγμή, θα δούμε πώς θα τις αξιολογήσουμε και βεβαίως είναι σημαντικό να υπάρχουν στη χώρα αυτή ε, δημοκρατικές σχέσεις. Ε, από ό,τι είδαμε, τέσσερα χρόνια μετά δεν έχει καθόλου βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με το πώς διεξάγονται οι εκλογές. Ευχαριστώ. Η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων δεν ξέρω ποιος. Είναι και ο Χωσέ Αντώνιο εδώ. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει το λόγο. Um, just um, a small comment. Ναι, ένα σύντομο σχόλιο. Ήταν πολύ πιο προβληματικές αυτές οι εκλογές σε σχέση με αυτές τις Σενεγάλης. Προφανώς, δεν χρειάζεται να σα το πω εγώ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τη Μαρία που άντεξε όλες αυτές τις ε, φάσεις της διαδικασίας. Ενδιαφέρον αυτό που είπατε για, τις, για την τεχνολογία και τις αποτυχίες και τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει. Αν θυμάστε πέρσι, είχαμε θίξει το θέμα αυτό στην ε, διάσκεψη εδώ στο Κοινοβούλιο υψηλού επίπεδου. Και στην ΕΙΕΔ προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε να το δουλεύουμε το θέμα αυτό. Έχουμε την ε, εντολή από τη, από διακήρυξη των αρχών για να μπορέσουμε να εκπονήσουμε κάποιες ε, ε, κατευθυντήρες γραμμές και θέλουμε να παρουσιάσουμε την αρχική δουλειά που έχουμε κάνει και τα ευρήματα φέτος στο καλοκαίρι ήδη από την διακήρυξη των αρχών. Να δώσω τώρα το λόγο και στον Αντώνιο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα να υπογραμμίσω και εγώ τα σχόλια που έγιναν. Έχουν υπάρξει όντω διάφορα προβλήματα. Ξέρετε ότι εμείς ε, παρέχουμε στήριξη για την παρατήρηση εκλογών, παρέχουμε τεχνική βοήθεια και συστάσεις. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλα τα προβλήματα που υπήρξαν. Και όπως συζητήθηκε και, στις, ε, και από ε, τους των ε, αποστολών, μία από τις βασικές συστάσεις είναι ότι ναι, σημειώνουμε τις επιτυχίες, τα επιτεύγματα, ας πούμε, την, εθνική, ε, την επιτυχία της Εθνικής Επιτροπής, της Εφορευτικής, που μπόρεσε έτσι λιγάκι να κατευνάσει τα πνεύματα, ε, κυρίως ό,τι αφορά τα, ε, τις συγκρούσεις που οδήγησαν στον θάνατο δύο ατόμων και κυρίως πρέπει να δούμε το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να, δι, να στηρίζουμε τα, τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη διεξαγωγή των εκλογών στην χώρα. Οπότε υπογραμμίζουμε τα καλά και βεβαίως ε, τονίζουμε το δικό μας ενδιαφέρον και περιμένουμε και τις ε, ε, παρατηρήσεις της Εφαρτικής Επιτροπής για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στις μελλοντικέ εκλογές. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Άλλος κανείς, η Μαρία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να παρακολουθούμε την εξέλιξη της χώρας αυτής γενικότερα στο δημοκρατικό επίπεδο. Γενικά πάντως είναι μια χώρα η οποία παρόλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και ασφαλεία στην περιοχή του Σαέλ και των προσφύγων, γιατί δεν μιλήσαμε και για τους εκτοπισμένους εντός της χώρας, αλλά υπάρχει και ε, μια πραγματική πρόκληση μετακινούμενων πληθυσμών που έχουν σχέση και με την ε, αναθέρμανση του κλίματος, αλλά και τις συγκρούσεις που περιέγραψα κτηνοτρόφων και αγροτών και όλα τα ζητήματα των φυσικών πόρων και ιδίως του πετρελαίου. Νομίζω ότι υπάρχει, όπως είπα, ένα σημαντικό διακύβευμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που οδηγεί στην ανάγκη να διατηρεί στενή επαφή με τους Νιγηριανούς και για το θέμα το δημοκρατικό αλλά και γενικότερα για ό,τι ε, μπορεί να έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους για το έργο σας. Δεν ήταν εύκολη η αποστολή αυτή, παρόλα αυτά πολύ σημαντική όπως είπε ο κύριος Φίσας σημαντική χώρα της Αφρικής αυτή και εύπορη χώρα και βέβαια πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Ας κλείσουμε τώρα τη συζήτηση αυτού του θέματος, του υπαριθμού 10, και να προχωρήσουμε στις συνεδρίες και κλεισμένων των θυρών και όποιος ε, ε, οφείλει να αποχωρήσει, να αποχωρήσει. Λίγα λεπτά για να ε, επιτρέψουμε να αποχωρήσουν.